Θέλω να καλωσορίσω και τους συναδέλφους από τις άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, τους δημοσιογράφους επίσης. Θα ήθελα επίσης να ζητήσω από τους φωτογράφους να πάρουν τις τελευταίες φωτογραφίες και να καθίσουν στις θέσεις τους για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Θα ήθελα όλοι να βρίσκονται στις θέσεις τους το ταχύτερο δυνατό και έρχονται και οι τελευταίοι συνάδελφοι. Ελπίζω για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την ακρόαση του υποψηφίου επιτρόπου για τα ενεργειακά θέματα. Θέλω να καλωσορίσω τον Γκίντερ Ότιγκερ, τον Πρωθυπουργό του Κρατηδίου της Βάδης Βιρτεμβέργης. <clears throat> όπως ξέρετε, όπως καταλαβαίνετε και από τον τίτλο του, είναι πολιτικός πρώτης γραμμής σε ένα κράτος μέλος. Καλώς ήρθατε κύριε Έτογκερ. Χαιρόμαστε για την ευκαιρία που έχουμε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας. Πρόκειται για το θέμα της ενεργειακής πολιτικής που είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα προσφυλές και σημαντικό στην Επιτροπή μας και φυσικά έχει αυξηθεί και η σημασία του για την σύνολη ευρωπαϊκή πολιτική και είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάντα αμφιλεγόμενο σε πολιτικό επίπεδο και μάλλον θα παραμείνει αμφιλεγόμενο. Ένα θέμα το οποίο πάρα πολύ πιθανόν θα κερδίσει όλο και περισσότερη σημασία γιατί οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά από την έγκριση της συνθήκης της Λισαβόνας θα αυξηθούν. Χαίρομαι λοιπόν που είσαστε όλοι εδώ παρόντες και βλέπω ότι είναι και ο κύριος Λάινεν από την Επιτροπή Περιβάλλοντος παρόν και ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος θέλει και αυτή να συμμετάσχει πλήρως σε αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Μπορώ λοιπόν να σας υπενθυμίσω ξεκινώντας και πάλι τους κανόνες. Για την ακρόαση νομίζω τα είπαμε και χθε, αλλά το βασικό είναι να μπορέσετε να τηρήσετε τον χρόνο ομιλία σας, ώστε να μπορέσουν και οι τελευταίοι ομιλητές να θέσουν τα ερωτήματά τους και σας παρακαλώ να έχετε κατανόηση ότι όταν δεν τηρείτε το χρόνο σας, και αυτό ισχύει για όλους, εγώ θα αναγκαστώ να σας διακόψω. Αυτό δεν το κάνω από κακοβουλία, Απλώ το κάνω για να προστατεύσω τα δικαιώματα όλων των βουλευτών να θέσουν ερωτήματα. Καλώ ήρθατε λοιπόν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Ετουγκέρ, ο οποίο έχει το λόγο για ένα διάστημα μέγιστο 10 λεπτών. Οι περισσότεροι συνάδελφοι σα γνωρίζουν και μπορείτε να παρουσιάσετε λοιπόν τα ζητήματα που σα ενδιαφέρουν. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία να έλθω ενώπιον της Επιτροπής Βιομηχανία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση και είναι μια ευκαιρία για να, να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή απόψεων. Όπως ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι εάν επικυρωθώ από το Κοινοβούλιο θα μπορέσω να συνεργαστώ μαζί σας στα πλαίσια μιας στενής εταιρικής σχέσης. Εμείς βρισκόμαστε σήμερα ενώπιον ενός νέου κεφαλαίου. Ενός νέου κεφαλαίου, το οποίο μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας, για πρώτη φορά ε, αντιμετωπίζεται μέσα από νέες δομές, ε, μέσα από νέες δομές και στην Κομισιόν και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που είναι εκλεγμένο και από δομές του Συμβουλίου και υπάρχουν σημαντικές προσδοκίες σε σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη της ε, πολιτικής ενέργειας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρισκόμαστε στο μέσο μιας χρηματοοικονομικής κρίσης και σε τοπικό επίπεδο και σε περιφερειακό επίπεδο και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν ληφθεί σημαντικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά δεν έχουμε περάσει ακόμα την κρίση, δεν την έχουμε ξεπεράσει. Αλλά η κρίση αυτή για την Ευρώπη, τα κράτη-μέλη της, για τους πολίτες της, δεν θα πρέπει <clears throat> να είναι μονάχα κάτι αντικό. Θα είναι και μια ευκαιρία να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο ασκούμε την πολιτική μας. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όπως το παρελθόν. Θα πρέπει να εργαστούμε πολύ περισσότερο από κοινού. Θα πρέπει να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί, να εξασφαλίσουμε και την αηφορία, να εξασφαλίσουμε την κοινωνική δικαιοσύνη επί τη βάση νέων κατευθύνσεων τις οποίες θα πρέπει να χαράξουμε. Αυτό ισχύει για όλες τις μορφές της οικονομικής πολιτικής, αλλά ακόμα περισσότερο και στην περιοχή της πολιτικής ενέργειας, όπου πρέπει να ανοίξουμε νέα κεφάλαια. Με την συνθήκη της Λισαβόνας και το άρθρο 194 έχουμε ένα νέο νομικό πλαίσιο, το οποίο για πρώτη φορά μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ευρείες νομικές αρμοδιότητες. Και ανοίγει το δρόμο για μια ευρωπαϊκοποίηση της ενεργειακής πολιτικής μέσω κοινών ε, κατευθύνσεων που θα χαράξουμε σε πλαίσιο νομοθετικό, που θα χαράξετε δηλαδή εσείς μαζί με το Συμβούλιο και είναι απαραίτητο να κτίσουμε πάνω σε αυτά τα οποία έχουν επιτευχθεί ήδη τα τελευταία πέντε χρόνια, τα σημαντικά μέτρα που έχουν ληφθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Πριν από δέκα χρόνια η ενέργεια δεν ήταν θέμα που απασχολούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από πέντε χρόνια μονάχα αρχίσαν οι πρωτοβουλίες στον τομέα αυτό. Αυτά τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια με κανονισμούς, με οδηγίες, με αποφάσεις, με προτάσεις, με πακέτα, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πιστεύω ότι τα επόμενα πέντε χρόνια, εάν με επικυρώσετε, θα μπορέσω να δώσω μια σημαντική συνεισφορά στην ευρωπαϊκοποίηση της ενεργειακής πολιτικής σε στενή συνεργασία με αυτά τα οποία γίνονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, δηλαδή με πλήρη σεβασμό της αρχής της επικουρικότητας. Εγώ γνωρίζω πολύ καλά την κοινοβουλευτική διαδικασία. Επί 14 χρόνια ήμουν βουλευτής σε τοπικό κοινοβούλιο. Εδώ και 26 χρόνια σχεδόν βρίσκομαι και σε τοπικό κοινοβούλιο στην χώρα μου. Έχω μια εμπειρία εδώ και πέντε χρόνια ως Πρωθυπουργό του κρατηδίου μου. Γνωρίζω λοιπόν τι, τι πρέπει να αναμένω από ένα κοινοβούλιο και από τους πολίτες. Υπάρχει μια σχέση εκτελεστικής εξουσίας με κοινοβουλευτική εξουσία που θα πρέπει όλοι μας να λάβουμε υπόψη μας και πιστεύω ότι θα είναι επωφελές για όλους μας να μπορέσουμε από κοινού να προωθήσουμε τα θέματα αυτά που άπτονται της πολιτικής ενέργειας. Τόνισε και πάλι ότι είναι εξ, εξέχουσας σημασίας η πολιτική ενέργειας και αφεαυτής και ως παράγον για την οικονομική ανάπτυξη και εξάλλου οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν τα αποτελέσματα μια ενισχυμένη εσωτερική αγορά και τέλο η ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο στην κλιματική αλλαγή και στην αηφορία. Με την ε, συνθήκη τη Λισαβόνα έχετε αποκτήσει σημαντικέ διευρυμένε <clears throat> αρμοδιότητε και εδώ ένα <clears throat> νέο κανόνα του παιχνιδιού είναι η αλληλεγγύη. Όλοι ανεξάρτητα από το πού προέρχεστε, θα πρέπει να έχετε την ε, ευαισθησία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον τομέα <clears throat> της ε, πολιτικής ενέργειας, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα σύνορα και τα όρια τα οποία τίθενται για μια συνολική ρύθμιση των θεμάτων αυτών. Εγώ είμαι έτοιμος να διερευνήσω λοιπόν όλα τα όρια τα οποία υπάρχουν για να προχωρήσουμε σε μια ω το δυνατόν πιο συνεκτική πολιτική. Είναι απαραίτητο να τορίσουμε την ανταγωνιστικότητα, όπως είπα, την αηφορία <clears throat> και κυρίως να εξασφαλίσουμε την τόσο σημαντική για την Ευρώπη ασφάλεια εφοδιασμού. Οι στόχοι του 2020 ε, είναι απαραίτητο να επιτευχθούν μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι στόχοι αυτοί οι οποίοι είναι φιλόδοξοι θα πρέπει να εξυπηρετηθούν με συγκεκριμένα βήματα τα οποία θα εξασφαλίσουν τους στόχους στους οποίους έχουμε θέσει. Και αυτό είναι, αυτό είναι το σημαντικότερο καθήκον μας. Η σημερινή πραγματικότητα <clears throat> είναι τέτοια που τα ορυκτά καύσιμα τα οποία αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στην ε, οικονομία μας, μας οδηγούν και σε εξάρτηση από εισαγωγές. Γι' αυτό το λόγο χρειαζόμαστε να προχωρήσουμε σε μια συνολική αλλαγή υποδείγματος στην πολιτική ενέργειας με το στόχο του να αποσυνδεθούμε από την οικονομία του άνθρακος, να έχουμε μια οικονομία φτωχή σε του άνθρακο και συγχρόνω να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού στην Ευρώπη και την αλληλεγγύη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο στόχο του 20% για την ενεργειακή απόδοση είναι ένα βασικό στοιχείο αυτή τη πολιτική που ακόμα δεν έχει επιτευχθεί. Θα πρέπει εμεί να παρακολουθήσουμε την πρόοδο και να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε περαιτέρω μέτρα, ώστε μέσα στα επόμενα χρόνια να μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και να μην παραμείνει μονάχα στα χαρτιά. Η... Το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από την επιτυχία με την οποία θα μπορέσουμε να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους που έχουμε θέσει στον τομέα της ενέργειας και που θα πείσουν και τον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος έχει ακόμα κάποιο σκεπτικισμό σε σχέση με την ικανότητα της Ευρώπης σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Γι' αυτό θα πρέπει να αναλύσουμε το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή απόδοση και επί τη βάση αυτού να προχωρήσουμε σε νέα εστιασμένα σχέδια για την περαιτέρω βελτίωση των στόχων μας. Η βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, της ασφάλειας εφοδιασμού, είναι ένας δεύτερος σημαντικός ρόλος για μας, που έχει μια διάσταση και εσωτερική στην Ευρώπη και μια εξωτερική διάσταση. Ό,τι αφορά κυρίως την εξωτερική πολιτική, πιστεύω ότι χρειάζεται να υπάρξει μια ε, μεγαλύτερη προσπάθεια σφυριλάτησης μιας κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής αντί του να βασιζόμαστε μονάχα σε διμερείς συμβάσεις και συμφωνίες <clears throat> για τον ενεργειακό τομέα. Και αυτό το λέω υπενθυμίζοντας και την δική μου <clears throat> ιδιαίτερη πατρίδα. Έχουμε διαπιστώσει ότι μόνο με την συνεργασία αυτή μπορούμε σε μακροχρόνιο επίπεδο να αποκομίσουμε τα ωφέλη τα οποία θέλουμε να έχουμε. Έχουμε, λόγω της οικονομικής κρίσης, αποφασίσει μια σειρά από σημαντικά μέτρα για την βελτίωση και των υποδομών στον τομέα της ενέργειας, για την, για την ε, εσωτερική αγορά. Είναι σημαντικό για τον καταναλωτή και για την βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού απαραίτητη, απαράγραπτη η βελτίωση της ε, υποδομής ενεργειών. Όπως υπάρχει η βελτίωση της κινητικότητας στους ε, δρόμους, στα, σε δρομικές γραμμές, εσωτερικούς υδάτινους δρόμους και στις τηλεπικοινωνίες, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια εξίσου μεγάλη κινητικότητα για την ικανότητα μεταφοράς των φορέων ενεργείας. Να υπάρξει λοιπόν και ικανότητα μεταφοράς, να υπάρξει και διαφάνεια και συγχρόνως να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού μέσω αυτών των οδών μεταφοράς της ενέργειας και φυσικά θα παίξουν στο εγχείρημα αυτό σημαντικό ρόλο και οι ανανεώσιμες ενέργειες. Το τρίτο πακέτο για την εσωτερική αγορά <clears throat> θα πρέπει να το εφαρμόσουμε όλοι μαζί με την βοήθειά σας και να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά τα οποία παραμένουν ακόμα στην, στις ρυθμίσεις που αφορούν την εσωτερική αγορά. Πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς ευρωπαϊκά δίκτυα ενεργείας και τα οποία θα δώσουν και στον καταναλωτή μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής, μεγαλύτερη δυνατότητα διαδραστικής σχέσης με τους παραγωγούς ενέργειας. τα ευφυή e e δίκτυα, η e ευφυής παραγωγή ενέργειας δεν πρέπει να παραμείνουν μονάχα συνθήματα, πρέπει να γίνουν πραγματικότητα μέσα στην Ευρώπη. Πρέπει να δείξουμε λοιπόν ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε και σε ανοιχτό διάλογο και σε άτυπο και σε επίσημο επίπεδο και φυσικά μέσα στο πλαίσιο αυτό θεωρώ ότι τα ερωτήματά σας και οι απόψεις που θα διατυπώσετε θα είναι ένα πολύ καλό σημείο αφετηρίας για να διαμορφώσουμε μια πολιτική ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια. Έχετε λοιπόν τις προσδοκίες σας από μένα. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ σε αυτές και θα ακούσω πολύ προσεκτικά τις απόψεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τιγκέρ. Ο κύριος Δαλκουάδρας είναι ο πρώτος που έχει το <coughs> λόγο για να θέσει ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μα, Κύριε Επίτροπε, υποψήφιε Επίτροπε, προφανώς σα εύχομαι κάθε επιτυχία. Γνώριζετε πολύ καλά κύριε υποψήφιε Επίτροπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τον στόχο του 20% ανανεωσίμων ενεργειών στο μείγμα ενεργειών του για το 2020. Γνωρίζετε όμως εξάλλου ότι αυτός ο στόχος δεν είναι επαρκής εάν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε τους πολιτικούς μας στόχους σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα, τη μείωση των εκπομπών θεωρητού αερίου του θερμοκηπίου και εξασφαλίζοντας την ασφάλεια εφοδιασμού. Γι' αυτό, ορισμένοι πιστεύουν ότι μεταξύ των διαφόρων πηγών ενεργείας θα πρέπει να θέσουμε προτεραιότητες, να κάνουμε επιλογές. Άλλοι πιστεύουν ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το ερώτημά μου είναι απλό και πιστεύω σαφές κύριε υποψήφιε επίτροπε. Υποστηρίζετε ή θα, ήσασταν, ή θα υποστηρίζετε να θεσπιστεί ένας ολοκληρωμένος στόχος για όλες τις μορφές ενέργειας χαμηλών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου στο μέλλον με συνολικό τρόπο. Στόχοι δηλαδή για όλες τις μορφές αυτές ενέργειας. Ευχαριστώ. Κύριε Το 20% είναι ένας φιλόδοξος στόχος. Από την μέχρι τώρα εμπειρία μου και από την ιδιαίτερη μου πατρίδα, τη Βάδη Βιντεμβέργη, Μπορώ να πω ότι στην πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας έχουμε φτάσει στο 9% και έχουμε καλύτερα ποσοστά από το μέσο όρο της Γερμανίας και, στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος είμαστε στο 14%. Σωστό πιστεύω και ευφιές ήταν να προσδοριστούν φιλόδοξοι στόχοι και να επαληθευτούν οι στόχοι αυτοί μέσα σε ένα ορατό χρονικό διάστημα για να εξεταστεί αν συνεχίζονται ή όχι. Πιστεύω ότι μακροπρόθεσμα χρειαζόμαστε ένα ποστό ανώτερο του 20%. Το πώς θα εφαρμοστεί αυτό, το πώς θα εξασφαλιστεί και το πώς θα προσδιοριστεί συγκεκριμένα το ενεργειακό μείγμα εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα που παρουσιάζει κάθε περιφέρεια. Είτε πρόκειται για αιωλική ενέργεια, είτε πρόκειται για θερμική ενέργεια, είτε πρόκειται για ηλιακή παλαιριακή ενέργεια υπάρχουν διαφορετικές δυνατότητες, πραγματικότητες και δεδομένα στις περιφέρειες Ευρώπης. Και εδώ η επικουρικότητα με τα εθνικά κοινοβούλια και τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και τους τοπικά αρμόδιους φορείς θα έχει πολύ μεγάλο ρόλο να διαδραματίσει ως προς τον προσδιορισμό αυτού του μείγματος. Από πλευράς μας εμείς μπορούμε να συμβάλλουμε ως εξής μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, τη βελτίωση των δομών μεταφορών μεταφοράς ενέργειας. Και θέλουμε να έχουμε υψηλά πρότυπα για την ε, παραγωγή των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τα αιωλικά πάρκα τα οποία αναπτύσσονται σε αρκετές περιοχές αλλά χρειάζονται περισσότερα και επίσης χρειάζεται για τις, τα μεγάλα μετροπολιτικά κέντρα το Ρήνο και Ρούρ, το, την περιοχή των Παρισίων χρειάζεται να βρούμε λύσεις διαφορετικές και εκεί οι ευρωπαϊκές ε, το, το καθήκον της ευρωπαϊκής διάστασης θα ήταν και να προσδιορίσει ε, ένα προφίλ, μια γενική δηλαδή περιγραφή και να επαληθεύσει την τήρησή της αλλά και να διαμορφώσει τα δίκτυα που θα επιτρέψουν την ε, λήψη των αποφάσεων και την εμπλοκή των ενδιαφερόμενων παραγόντων στην υπόθεση αυτή. Για συμπληρωματική ερώτηση, κ. Φαλκουάντρας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έτιγκερ για την απάντησή σας. Αυτό το οποίο ήθελα να αναφέρω, όπως θα καταλάβατε κι εσείς, είναι στρατηγικές όπως αυτές οι οποίες λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο, <clears throat> όπου το μεγαλύτερο γνωστό σχέδιο για θαλάσσιες, θαλάσσια αιωλικά πάρκα, το οποίο θα φτάσει τα 32 γιγαβάτ το 2020, συνοδεύεται από μία αναζωγόνηση του προγράμματος πυρηνικής ενεργείας. Αποσχάσει. Δηλαδή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο λαμβάνει υπόψη όλες τις πηγές χαμηλών εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Αυτό ήταν το ερώτημά μου λοιπόν αν κύριε Επίτροπε εσείς θα υποστηρίζατε μια τέτοια προσέγγιση. <clears throat> δηλαδή να προωθήσουμε συγχρόνως όλες τις πηγές ενέργειας που οδηγούν σε χαμηλή εκπομπή αερίου του θερμοκηπίου και όχι μονάχα ένα τμήμα Πρόεδρος. Αγαπητοί συνάδελφοι, εχθέ ε, καταφέραμε να τηρήσουμε σχεδόν χωρί ε, δυσκολία τον χρόνο μα. Σήμερα βλέπω ότι είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό παρακαλώ να είμαστε αυστηροί. Ένα λεπτό ερώτηση, δύο λεπτά απάντηση, μισό λεπτό ε, συμπληρωματική ερώτηση, ένα λεπτό απάντηση για να μην χάσουμε τον χρόνο μα. Παρακαλώ. Κύριε Ότιγκεν. Η μέση οδός από τα όσα προτείνετε εσείς νομίζω ότι είναι η ορθότερη. Να έχουμε ένα περιθώριο δηλαδή και για την λειτουργία της ε, οικονομίας και των εθνικών οργάνων, αλλά και συγκεκριμένα καθήκοντα που θα πρέπει να προσδιοριστούν από το δικό μας επίπεδο. Και ουσιαστικά μπορούμε να βρούμε έτσι το δρόμο από μία η οικονομία που έχει πολύ ψηλέ εκπομπέ του οξυδίου του άνθρακα σε μια οικονομία που είναι απαλλαγμένη θα έχει χαμηλέ εκπομπέ του οξυδίου του άνθρακα. Εδώ εγώ τρεφώ κάθε ε, σεβασμό για τι εθνικέ διαδικασίε λήψεων αποφάσεων και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη Βάδη Βερτεμβέργη έχει ε, και εκείνη τη συμβολή της στον εθνικό, εθνικό μηχανισμό λήψη αποφάσεων και για τα πυρηνικά οργοστάσια και την απόφαση για την παράταση της ζωής τους, ε, της λειτουργίας τους. Εδώ οι εθνικές αρμοδιότητες, οι τοπικέ αρμοδιότητε νομίζω πρέπει να τύχουν κάθε σεβασμού. Είναι ζήτημα εθνικών κυβερνήσεων και τοπικών εθνικών πληθυσμών το να κρίνουν αν θέλουν τα πυρηνικά ή όχι. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Αυστρία έχουν, πάρει τις, έχουν κάνει τι επιλογέ του. Υπάρχουν άλλες χώρες ε, οι οποίες μπορεί να θεωρούν ε, την ε, λύση αυτή προσωρινή, κάποιες άλλες που τη θεωρούν μακροπρόθεσμη, κάποιες που να μην τη θέλουν καθόλου. Και γι' αυτό πρέπει να σεβαστούμε τις διαφορετικές επιλογές του καθενός. Από την άλλη και η έρευνα και οι ψηλές προδιαγραφές θα πρέπει να αποτελέσουν επίκεντρο των εργασιών μας στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Έτσιγκερ δική μου ερώτηση δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με την ενεργειακή πολιτική, αλλά με τη γενικότερη στάση που θα έχουμε απέναντι στι ε, πολιτικέ επιλογέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν στη Βάδη Βιτεβέργη, ε, και σε εσά συγκεκριμένα ως Πρωθυπουργού έχουν εκφραστεί επικρίσεις στο τελευταίο διάστημα ε, ως προς την οικονομική, τις οικονομικές επιλογές. Τι θέλει λοιπόν για μένα το ερώτημα πώς μπορείτε με τα νέα καθήκοντα που θέλετε να αναλάβετε να ε, διαχειριστείτε ζητήματα που έχουν να κάνουν με 27 κράτη-μέλη εάν ε, δεν ήσταν σε θέση να τηρήσετε ευρωπαϊκές προδιαγραφές ε, στα οικονομικά θέματα μέσα σε ένα κρατήδιο της Γερμανίας. Ο κύριος Φαν Απάντηση. Όχι. Δεν υπάρχει ζήτημα εδώ. Υπάρχει, ένα, ε, υπάρχει μια αρχή σχετική με, ε, την κατανομή των χαρτοφυλακίων, ποιο είναι υπεύθυνο στο περιφερειακό επίπεδο, στο ομοσπονδιακό επίπεδο, ποιο είναι στο ομόσπονδο επίπεδο υπεύθυνο. Και του 17 ε, μήνες που είχα εγώ την διακυβέρνηση του κρατηδίου, τηρήσαμε τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού δικαίου και ο Υπουργός των Εσωτερικών του κρατηδίου μας στήρισε απολύτως τα, ε, τις διατάξεις σχετικέ με την πάταξη της νομοποίησης παράνομων εσόδων. Επέβαλε μάλλον την αυστηρή των διατάξεων αυτών. Φάνηκε εντωμεταξύ ότι οι προδιαγραφές αυτές ε, είχαν προχωρήσει όπως έπρεπε από το Προεδρείο της κυβέρνησης, δηλαδή μια ενδιάμεση αρχή, ε, σε ε, αυστηρή τήρηση παρά τις κατηγορίες που είχαν διατυπωθεί και ότι τελικά τηρήθηκαν όπως έπρεπε οι προδιαγραφές αυτές για την ε, αντιμετώπιση της νομοποίησης παρανόμων εσόδων. Και πρέπει να σα πω ότι ούτε καν το δικό σα κρατήριο, ούτε κανένα άλλο στη Γερμανία είχε τόσο αυστηρό έλεγχο όσο η Βάδη Βιρεμπέργη. Δευτερεύους ε, συμπληρωματική ερώτηση ο κύριο Γκλάντε. Εντάξει, εμείς βέβαια δεν έχουμε και καζίνα στην, ε, στο Βραδεμβούργο. Ίσως αυτό είναι το θύμα. Για την ενεργειακή πολιτική. Πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε με τον κύριο Μπαρός ώστε να εξασφαλίσετε περισσότερη έρευνα για την ενέργεια που είναι απαραίτητη πιστεύω. Κύριος Φενότσιγκερ, αγαπητοί συνάδελφε, νομίζω ότι εδώ το χαρτοφυλάκιο αυτό θα πρέπει να διονγκωθεί, να μεγαλώσει σιγά σιγά, όπω άλλωστε έχει γίνει ήδη στο παρελθόν με τον προκάτοχό μου, όπω άλλωστε έχουν, έχει γίνει και με το δικό σα χαρτοφυλάκιο, με τι εξουσίε και αρμοδιότητε τη δική σα ε, ε, επιτροπή, γιατί έτσι πρέπει να γίνει και είμαι αποφασισμένος το χαρτοφυλάκιό μου να το καταστήσω αποτελεσματικό και ουσιαστικό. Βεβαίως υπάρχουν όρια, τα όρια τα οποία ορίζει κάθε δημοκρατική αρχή για κάθε δημοκρατικό ε, όργανο. Φερρυπίν, περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, έρευνα, ιστορική αγορά, ανταγωνισμός, οικονομία, εξωτερική πολιτική. Ο συλλογικό όργανο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βέβαιος ότι θα μπορέσει με εταιρικό πνεύμα και με αμοιβαία, σε αμοιβαίο πνεύμα συνεργασία και όχι σε ε, αποκομμένες προσπάθειες ε, διαμόρφωσης πολιτικών να προωθήσει την έρευνα και με το προσδιορισμό των ε, αρμοδιοτήτων όπως γίνεται, όπως πρέπει να γίνεται, εγώ θα έχω την αρμοδιότητα και για την έρευνα για την ενέργεια. Είναι ένα καθήκον το οποίο με σοβαρότητα θα επιτελέσω και σε συνεργασία βεβαίως με τους συναδέλφους που θα έχουν αντίστοιχες συγγενείς αρμοδιότητες, αλλά πάντως σε σεβασμό των ορίων της κατανομής των αρμοδιοτήτων αυτών. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Έκ έχει το λόγο. Η κυρία Έκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. παρά το γεγονός ότι υπήρξε αυτό το πακέτο για την ενεργειακή αγορά, το τρίτο πακέτο λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι η εσωτερική αγορά δεν λειτουργεί ακόμα πλήρως στον τομέα της ενέργειας. Οι καταναλωτές και η βιομηχανία αντιμετωπίζουν προβλήματα σε ό,τι αφορά την ε, μεταφορά μέσω των δικτύων, μέσω των ε, διακοιμάσεων των τιμών, μέσω των προβλημάτων από την κλιματική αλλαγή και η Ευρώπη δεν έχει επιτύχει ουσιαστικά τίποτα σε ό,τι αφορά την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Γι' αυτό είναι απαραίτητε νέες αποφάσεις με ταχύ ρυθμό και σημαντικές ενέργειες οι οποίες θα οδηγήσουν στη, στη λύση αυτών των προβλημάτων. Αυτά τα οποία αναφέρονται λοιπόν στο στο Συμβούλιο τι μέτρα εσείς θέλετε να προτείνετε να προχωρήσουν, να προ... θα, θα, θα, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτά με γρήγορο τρόπο. Κύριε Έτουγκερ, έχετε το λόγο. Κυρία Εκ, θα ήθελα καταρχήν να τονίσω ότι η πλήρης εφαρμογή του τρίτου πακέτου για την ενεργειακή αγορά θα πρέπει να εξασφαλιστεί, θα πρέπει να τύχει ελέγχου και επίσης μαζί σας θα πρέπει να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Πρώτα απ' όλα, πρόκειται για το δεκαετές σχέδιο επενδύσεως των επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον τομέα του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος. Πρέπει να πείσουμε τις βιομηχανίες και τους φορείς ενέργειας να βελτιώσουν την ικανότητα μεταφοράς των δικτύων τους μέσα στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη επίσης τα επιμέρους ε, δίκτυα σύνδεσης, είτε είναι βόρεια-νότια είτε ανατολικά-δυτικά, θα πρέπει να ενισχυθούν ακολουθώντας το παράδειγμα του ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου. Όπως είχαμε τα διευρωπαϊκά δίκτυα για το σιδηρόδρομο, θα πρέπει να γίνει κάτι αντίστοιχο για τις ε, διασυνδέσεις ηλεκτρικών δικτύων, ώστε να υπάρχει η πλήρης αυτή δυνατότητα να είναι διασυνδεδεμένες όλες οι γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού ε, αερίου και να έχουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο. Αυτό φυσικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και στις ε, συζητήσεις για τον προϋπολογισμό τα επόμενα χρόνια και να προετοιμαστούν οι απαραίτητες λύσεις. Δεύτερον, κατά την άποψή μου, είναι απαραίτητο να υπάρχει πληρέστερη πληροφόρηση προ του καταναλωτέ στα πλαίσια τη εσωτερική αγορά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να ενισχυθεί ο καταναλωτή έναντι των επιχειρήσεων με το να έχει καλύτερε γνώσει σε σχέση με τι δημόσιε πρωτοβουλίε, με τα μέσα τα οποία είναι στην διάθεσή του, με τι νέε ε, δυνατότητες οι οποίες ανοίγονται με καλύτερη κατάρτιση και εκπαίδευση νομίζω ότι όλα αυτά είναι απαραίτητα για μια καλύτερη γνώση από την πλευρά του καταναλωτή. Τρίτον, θα πρέπει ο καταναλωτής να μπορεί να χρησιμοποιήσει με ενεργό τρόπο αυτές τις πληροφορίες που θα αποκομίσει. Δηλαδή να υπάρχει μια διαδραστικότητα ώστε να μπορεί να γνωρίζει ο καταναλωτής και πού θα μπορεί να βρει φθηνότερο φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι ένα αποφασιστικό θέμα και είναι πάρα πολύ σημαντική και η λεγόμενη αποδεσμοποίηση, το unbundling. Υπάρχει μια συζήτηση η οποία είχε γίνει στο παρελθόν για τα θέματα αυτά και η οποία υπήρξε μια αμφιλεγόμενη συζήτηση με επιχειρήματα υπέρ και κατά γνωρίζω ποια είναι, ποιες είναι οι απόψεις μέσα στη δική μου κυβέρνηση, μέσα στη δική μου χώρα, αλλά το θέμα της επίσημης μεταφοράς της πώληση των δικτύων για μένα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από πλήρη διαφάνεια. Το να επιτύχουμε λοιπόν την πλήρη διαφάνεια σε σχέση με την ιδιοκτησία των δικτύων είναι απαραίτητο. Κύριε Έτιγκερ, σας παρακαλώ πάρα πολύ να παραμείνετε μέσα στα πλαίσια του χρόνου σας. Κυρία Έκαρτ. Ε, ε, Κύριε Έτιγκερ, τα μέτρα τα οποία αναφέρατε, αυτά απαιτούν κάποιο χρόνο. πρέπει να υπάρξει μια βελτίωση των δομών της βιομηχανίας, θα πρέπει να πληροφορηθεί καλύτερα ο καταναλωτής. Όλα αυτά χρειάζονται πολύ χρόνο. 50% των ενεργειακών μας αναγκών στην Ευρώπη καλύπτονται από εισαγωγές. Και το 2020 μπορεί αυτό να φτάσει το 70%. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω από εσά τι έχετε να προτείνετε ήδη πριν από την Νεαρινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε σχέση με την ενεργειακή ε, απόδοση. Κύριε Έτιγκερ. έχω τονίσει ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα σημαντικό στοιχείο και η Ισπανική Προεδρία κινείται προς την ίδια κατεύθυνση. Μετά από την Κοπενχάγη είναι σαφές ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε σημαντικά την ενεργειακή απόδοση. Θα χρησιμοποιήσω τις επόμενες εβδομάδες για να μπορέσω και μαζί σας να παρουσιάσω συγκεκριμένες προτάσεις για τα θέματα αυτά και σε συμφωνία με την κυρία Χέντεγκάρτ και με όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στον τομέα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής να μπορέσουμε να δώσουμε τις απαραίτητες κατευθύνσεις για μια τέτοια ενεργειακή πολιτική. Ευχαριστώ κύριο Στούρμες. Κύριε Έτεγκεν, καλώ ήρθατε σε αυτή την ακρόση. Μια ισχυρή ενεργειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση με φιλοδοξίε αφορά το να μιλάμε με μια φωνή στη Ρωσία. στι γερμανικέ εφημερίδε φέρεστε ότι είπατε ότι ένα κομμάτι των καθηκόντων σας είναι να επερασπιστείτε τα γερμανικά συμφέροντα. Πώς ταιριάζουν αυτά. Αναφέρατε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντα ήταν να, να πολεμά για το, για το διαχωρισμό ιδιοκτησίας, το ownership unbundling. Αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση που είναι πιο κοντά στα συμφέροντα των μεγάλων γερμανικών εταιριών. Αλλά η μεγαλύτερη πολιτική σα μάχη τα επόμενα χρόνια θα ήταν να επιβάλλετε φιλόδοξε πολιτικέ ενεργειακή απόδοση Είσαστε έτοιμος να πολεμήσετε για 20% στόχο δεσμευτικό για αποδοτικότητα της ενέργειας και ε, να, αλλάξουν η να αλλάξει η οδηγία για την ΚΑΠ και να αλλάξει η οδηγία για ενεργειακές υπηρεσίες. Διότι η πολιτική και η ενεργειακή απόδοση είναι αυτό που πρέπει να εφαρμόσετε επόμενα χρόνια. Και αν αυτό όμως συγκρούεται με τα συμφέροντα των μεγάλων γερμανικών ε, λιγοπολίων, πώς θα αντιμετωπίσετε το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Σαφής η ερώτηση, κύριε Έτσιγκερ. Κύριε Τσούρμες. Για μένα είναι δεσμευτικά τα όσα έχουν ήδη συμφωνηθεί. Και 20% και όλα αυτά τα οποία ε, ήδη έχουν ε, προσδιοριστεί, έχουν ήδη κρυθεί και από εσά τους ίδιου και από του προκατόχους μου, ασφαλώς με δεσμεύουν. Καθήκον μου, εν προκειμένου θα είναι μετά το 2020 να δούμε τι θα γίνει και το 2050 μακροπρόθεσμος στόχος δηλαδή, να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε την απαλλαγή από τον άνθρακα. Δηλαδή τη μεθεπόμενη δεκαετία θα πρέπει να συζητήσουμε πώς θα αναπτύξουμε, θα ορίσουμε και θα επιτελέσουμε στόχους. Είναι ήδη δεδομένες οι πρωτοβουλίες για τον διαχωρισμό είναι γνωστές. Αλλά το πώς θα γίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, η διαφάνεια δηλαδή πώς θα εξασφαλιστεί, η ε, σχέση ε, κόστους και ωφέλους, η λειτουργία του συστήματος αυτού θα πρέπει να προσδοριστούν στην συνέχεια. Χώρες όπως η Γερμανία και η Γαλλία που είναι μεγάλη παραγωγή και καταναλωτές ενέργειας θα πρέπει να μπουν στο μικροσκόπιο για να τηρηθούν όλες τις συνθήκες ε, αντικειμενικότητας. Επίτροπος της Γερμανίας, ως υποψήφιος επίτροπος από πλευράς Γερμανίας εκτίθαμε ενώπιον σας, αλλά θα είμαι Ευρωπαίος Επίτροπος, Ευρωπαϊκός Επίτροπος. Δεν θα είμαι δηλαδή μεροληπτικός υπέρ της Γερμανίας των γερμανικών δομών. Και ενώπιον σας και σε θέματα ακόμη οικονομικά, αλλά σε κάθε άλλο τομέα θα έρχομαι για να υποστηρίξω τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Ο κύριος Τούρμας έχει τίποτα άλλο να συμπληρώσει. Uh, λοιπόν, είναι ανοιχτό μυστικό ότι έχετε στενές προσωπικές σχέσεις και τον κύριο Μπένουτ Χάρτ που είναι πρόεδρος της ΙΟΝ και τον κύριο Γκρόσμαν πρόεδρο της AWE, της AWE. Πώς ασχολείστε με θέματα της διαμαρτυρίας της WWF κατά του συστήματος αδειοδότησης για το, τη μονάδα παραγωγής που χρησιμοποιεί άνθρακα στην Καλσούη και πώς θα ξεκινήσετε ενδεχόμενες ε, ε, διαδικασίες παράβασης κατά της Άμπλιον που, που δεν, έχει προβεί, δεν ανήκει στο κομμάτι που έχει αποσυνδεθεί της AWE δεν αμφισβητώ ότι διαγράφετε όποιον θέλετε, ότι... Αλλά πρέπει να έχετε διαβεβαιώσεις λοιπόν ότι η πολιτική δεν αποφασίζεται εκεί τελικά, ότι παίρνετε εσεί τις αποφάσεις. Ε- Κύριε Τσίγκερ, σας παρακαλώ να ε, πιστέψετε ότι θα έχω την απαραίτητη αντικειμενικότητα, αμεροληψία και διαφάνεια που χρειάζεται σε αυτή την θέση και που είναι απαραίτητη σε μια δημοκρατία. Ναι. Παίξαμε με τον κύριο αυτών ε, τη ΣΟΕ για ε, ένα ε, γκαλά, για ένα φιλανθρωπικό ουσιαστικά αγώνα και μάλιστα δεν ήταν και πολύ καλός παίχτης πρέπει να σας πω. εάν αυτό συνέβαλε στον φιλανθρωπικό μας σκοπό, γιατί όχι. Παίξαμε επίσης σε μια άλλη αίθουσα ταυτόχρονα στο, στο χώρο των εγκαταστάσεων, στις εγκαταστάσεις μας, αλλά δεν έπαιξα εγώ μαζί του, εκείνος έπαιζε με και εγώ με άλλους. Το θέμα όμως είναι ότι μου φέρε χρήματα εκεί που τα χρειαζόμουν για να τα διαθέσω όπως ε, ήταν σκοπιμά τώρα. κύριος Τσίτσεστερ, επόμενη ερώτηση. Mr. Ettinger, bearing in mind... Κύριε Έτιγκερ, λαμβάνοντα όψη ότι 31% περίπου της ευρωπαϊκής ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από πυρηνική ενέργεια, Νομίζετε ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα αυτό το στοιχείο να αντικατασταθεί από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ακόμα και με έργα μεγάλης ε, ε, προγράμματα όπως Desert Tech, όπως ηλιακά, στη Σαχάρα ε, ή ακόμα και με μεγάλα φράγματα. Και σε αυτό το πλαίσιο Πιστεύετε ότι μπορείτε να λάβετε μεγάλες πρωτοβουλίες, μεγάλα προγράμματα κατά τη θητείας σας ή θα εστιαστείτε στο να χρησιμοποιείτε το πακέτο, το πακέτο για το κλίμα υφιστάμενη νομοθεσία πλήρως εκτελέσιμα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ κύριε Έτσιγκερ. Το πακέτο για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει να επιτευχθεί πλήρως. Είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο και είναι απαραίτητο να ε, εκπληρωθεί γιατί παίζει και σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά την ακτινοβολία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλο τον κόσμο. Εγώ θεωρώ λοιπόν αυτούς τους στόχους ότι είναι σημαντικοί και ορθοί. Εμείς τον επόμενο χρόνο θα πρέπει να αποφασίσουμε τι θα πράξουμε την επόμενη δεκαετία. Και θα πρέπει επίσης να αποφασίσουμε πού και πότε μπορούμε να θέσουμε περαιτέρω στόχους σε τεχνικό ε, επίπεδο και σε επίπεδο υλοποίησης πέραν του 2020, κατά την άποψή μου. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, οράματα και σχέδια όπως το Desert Tech με όλους τους εμπλεκομένους. Είναι ένα θαυμάσιο σχέδιο, μια θαυμάσια ευκαιριακή για την Αφρική και για την Ευρώπη. Η ηλιακή ενέργεια λοιπόν μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο για όλους μας και μπορεί επίσης να προωθήσει την δημιουργία δικτύων μεταφοράς ενέργειας τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Δηλαδή δίκτυα μεταφοράς ενέργειας τα οποία να έχουν πολύ χαμηλό ποσοστό απώλειας ενέργειας. Είναι λοιπόν κάτι στο οποίο πιστεύω ότι θα πρέπει να προσκαλέσουμε όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο της παραγωγής ενέργειας και μεταφοράς ενέργειας να λάβουν μέρος σε αυτό επίσης αυτούς οι οποίοι εργάζονται στον τομέα των επικοινωνιών. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μια εκμετάλλευση της Αφρικής. Θα πρέπει να οδηγήσει σε μια νέα εταιρική σχέση με την Αφρική σε, στα πλαίσια μιας εταιρική σχέσης win-win προς αμοιβαίο όφελος για να μπορέσει λοιπόν να εξασφαλίσει και την γεφύρωση των δύο πλευρών της Μεσογείου. Σε ό,τι αφορά την πυρηνική ενέργεια υπάρχουν χώρε στις οποίες θα παίξει σημαντικό ρόλο η πυρηνική ενέργεια και την επόμενη δεκαετία, Όπω είναι και η Γερμανία. Υπάρχουν άλλες χώρες οι οποίε για την ε, πυρηνική ενέργεια βλέπουν αυτή την ενέργεια όχι μόνο σαν μια τεχνολογία γεφύρωση, αλλά ω μια τεχνολογία που θα μπορέσει να διατηρηθεί και στο διηνεκέ. Πρέπει να το δεχτούμε αυτό διότι παραμένει η απόφαση αυτή για το ενεργειακό μείγμα απόφαση των εθνικών αρχών. Εγώ θα πρέπει να τηρήσω τα υπεσχημένα, να τηρήσω τις συμφωνίες οι οποίες έχουν συναυθεί. Συμπληρωματικό ερώτημα του κυρίου Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Στα αρχικά σας σχόλια, αρχικές παρατηρήσεις αναφερθήκατε ότι θα προσπαθήσετε να καλύψετε δίποτε κενά στο τρίτο πακέτο. Και εγώ παίξα ρόλο στη δημιουργία τη υπηρεσία για την συνεργασία των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών και έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν, πιστεύω. Εσεί θα υποστηρίξετε ενεργά το έργο του και ιδιαίτερα τι προσπάθειέ του για την επίλυση του θέματο ε, της αποσύνση ιδιοκτησία ή ownership on bundling. Σας ευχαριστώ. Κύριε Οι κανονισμοί αυτοί είναι, αποτελεσμα... αποφασιστική για να έχουμε μια πλήρη εσωτερική αγορά. Θα πρέπει να βρούμε τον μέσο δρόμο μεταξύ υπερβολικής ρύθμισης από τη μία πλευρά και από την άλλη μεριά μεταξύ μειωμένης ρύθμισης η οποία δεν έχει αποτέλεσμα στην αγορά. Οι ίδιες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η δική μου χρειάζεται να καλυφθούν από ρυθμίσεις οι οποίες θα είναι δίκαιες και οι οποίες θα οδηγούν σε πλήρη ανταγωνισμό. Επομένως θα πρέπει να αποφασίσουμε το ερώτημα του πώς βλέπουμε την ε, διαδικασία της, ε, της ρύθμισης σε περίπτωση που γίνεται κατά κάποιο τρόπο ε, κατάργηση ορισμένων εργοστασίων παραγωγής ενέργειας με κρατικές χρηματοδοτήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς γίνεται η δυνατότητα να πολιθούν ορισμένα από, αυτά τα, από αυτές τις ενεργειακές δομές και μέσα σε ποιο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία. Δεν έχει συμφωνηθεί αυτό ακόμα από όλα τα εθνικά κράτη πώς θα γίνει αυτό. Γι' αυτό ο φορέας που αναφέρατε νομίζω ότι μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στο να εξασφαλίσει τον καταλογισμό του πλήρους κόστους, την διαφάνεια, ώστε να υπάρξει μια σωστή αποτίμηση της αξίας αυτών των ε, εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και των πόρων ενέργειας. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ματίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι εδώ στα δεξιά σας. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, μιλήσατε πολύ για τα εργαλεία, για την πολυπικιλία των προτάσεων που έχουν τεθεί, τα διάφορα ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ένα από τα θέματα τα οποία αντιμετωπίσατε είναι ότι υπάρχει μια σειρά από ελλείψεις στον τομέα της ενέργειας και έχουμε αναφερθεί στην ανάγκη με περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Γι' αυτό θέλω να θέσω το εξής ερώτημα, το οποίο έχει ακριβώς να κάνει με το γεγονός ότι μέχρι στιγμής οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ενέργειας από την βιομάζα ήταν μέχρι στιγμής ιδιαίτερα άταλμες κατά την άποψή μου. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψή σας για το θέμα αυτό αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της ε, αποψήλωσης των δασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ξέρω αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προτείνει κάποιες δεσμευτικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της παραγωγής από βιομάζα. Um Σας παρακαλώ να λάβετε το λόγο για την απάντηση, κύριε Έτσιγκερ. Η βιοενέργεια ως θέμα είτε έχει να κάνει με τις μεταφορές, είτε έχει να κάνει με τη βιομάζα, πρέπει τα προσεχή χρόνια να εξεταστεί με πολύ ευαίσθητο και διαφοροποιημένο τρόπο και να αναπτυχθεί. Το 10% ως ποσοστό για τον τομέα των μεταφορών, παραδείγματι, είναι σχετικά αυστηρό όριο. Την οποία θα, το οποίο ποσοστό θα το τηρήσω απαράβατα, αλλά ε, σε σχέση και με τα ζητήματα που σχετίζονται με την ενέργεια. Δηλαδή θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσον αξίζει τον κόπο να ε, δούμε διαφορετική χρήση των οικολογικών επιφανείων, εκτάσεων, δηλαδή δασών κτλ. για να εξασφαλίσουμε μία αεφόρο πανεγωγή βιομάζας. Μια αεφορο παραγωγη δηλαδή, ένας οικολογικός και οικονομικός συνάμα απολογισμός πρέπει να γίνει ώστε να μην εξετάζουμε τη βιομάζα μεμονωμένα, πρέπει να κοιτάξουμε συνολικά τις συνέπειες ως προς τα ποσοστά εκπομπών σε διοξίδιο του άνθρακα. Το ίδιο και για τις ευαισθησίες ως προς τα τρόφιμα την στάση μας απέναντι στα τρόφιμα, απέναντι στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ευρώπη, επί παραδείγματι και την προοπτική τους. Είναι ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου, που θα πρέπει ε, ανάλογα με το πόσο θετικά συμβάλλουν στην, ε, στο συνολικό αυτό απολογισμό να προωθηθούν. Η κυρία Ματίας έχει συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε το ερώτημά μου έχει να κάνει με το στόχο της απόσυρσης από την χρήση άνθρακα και επειδή έχετε αναφέρει αυτό το ερώτημα θα ήθελα να σας ρωτήσω αν λαμβάνετε αυτός ο στόχος υπόψη στην πολιτική των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς θα θεσπίσετε πολιτικές οι οποίες λαμβάνουν υπόψη και τις ζημίες που παράγουν τα ορυκτά καύσιμα σε ό,τι αφορά την απερίμωση και την καταστροφή των εδαφών. Αν είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρχει μια πιο σαφής παρέμβαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Κυρία Έτυγγερ. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να εξετάσουμε και τις εισαγωγέ βιομάζας, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος σε τρίτα κράτη και ιδίω αναδυόμενα και αναπτυσσόμενα κράτη να ε, μην υπάρχει η επαρκής ευαισθητοποίηση. Εκεί πρέπει να δώσουμε έμφαση και με τα κίνητρα που θα προσφέρουμε και με τις δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς και με τα ποσοστά ή τα όρια που θα ορίσουμε για την συμμετοχή στον απολογισμό μας της βιομάζας της, προ... της προερχόμενης από τρίτα κράτη, αναδυόμενα ή αναπτυσσόμενα. Και τη συμβολή αυτής, υπολογισμό, δηλαδή στον, απολογισμό αυτών, στον ισολογισμό αυτών, της ε, συμβολής αυτής της βιομάζας στο, ε, ε στις εκπομπές του του άνθρακα. Σε αυτό είμαι διατεθειμένο να κάνω, καταβάλω ιδέες προσπάθειε. Διαφορετικά το αποτέλεσμα θα είναι ακριβώ το αντίθετο από το επιδιωκόμενο. Ευχαριστώ, κύριο Σάβάλλο. Κυρία Ζαβέλα. Τζαβέλα, με συγχωρείτε. Ότι και εκ μέρους της ε, ομάδος μου σας καλωσορίζω σε αυτή την ακρόαση και εύχομαι καλή επιτυχία στις επιδιώξεις σας. κύριε Άτικερ, μέχρι τώρα οι κανονισμοί, η νομοθεσία, η πολιτική και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλύπτουν το αέριο το οποίο προμηθευόμαστε μέσω κυρίως αγωγών έχετε την πρόθεση να παρουσιάσετε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη μεταφορά, την υγροποίηση και την νομική προστασία του LNG. Ευχαριστώ. Κύριε, Αυτό είναι ένα σημαντικό προϊόν από τις ε, πρώτες ύλες για οποιαδήποτε βιομηχανική χώρα και παίζει ακόμα σημαντικό ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα θέλω να συνεισφέρω το φυσικό αέριο να παράγεται κάτω από τις πιο αποδοτικούς δυνατόν όρους και η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει και στην περίπτωση του φυσικού αερίου εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης. Από το σχέδιο Nord Stream έχω τονίσει ότι είναι απαραίτητο να ισχύει το, το, η αρχή της ε, αλληλεγγύης και θα πρέπει να αντλήσουμε τα απαραίτητα διδάγματα για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξάλλου θα πρέπει να μειώσουμε την εξάρτηση είτε από, μία, από ένα διάβλο είτε από μία χώρα παραγωγής ε, φυσικού αερίου. Αυτό αφορά και τα δίκτυα μεταφοράς από την ε, Βαλτική και αυτά που έρχονται από την Ανατολική και Νότια Ευρώπη και από τα δίκτυα τα οποία έρχονται από τη Μεσόγειο, από την Αφρική παραδείγματος χάρη. Και εδώ θα πρέπει να λάβουμε και το θέμα της διασύνδεσης μέσα στην Ευρώπη, δηλαδή της κατανομής του φυσικού αερίου μεταξύ των χωρών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως όλα αυτά τα σχέδια θα πρέπει να αποφασιστούν μέσα στα επόμενα χρόνια. Θέλετε να θέσετε ένα συμπληρωματικό ερώτημα, κυρία Τζαβέλα. Εναλλακτικέ μορφέ ενέργεια. Τη Δευτέρα στο Στρασβούργο έχουμε την ακρόαση του υποψηφίου Επιτρόπου Βιομηχανία, κύριε Ότικερ, για να στηριχθεί η ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή επιχείρηση. Προτίθεστε να προωθήσετε ενεργειακή πολιτική που θα λαμβάνει υπόψη τα fuel mix που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενέργεια διαδραματίζει τεράστιο ρόλο στην ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην διασφάλιση θέσεων εργασίας. Όλο και αυξανόμενο μάλιστα ρόλο. Και για την ε, βιομηχανία των τροφίμων και για τη χημική βιομηχανία και για την παραγωγή ενέργειας, αλλά και για την διασφάλιση της, του εφοδιασμού σε ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει στρεφόμενοι κοιτώντας και τους άλλους μεγάλους παραγωγούς καταναλωτές, Ηνωμένε Πολιτείες, Ασία κτλ, να προωθήσουμε περισσότερο τις δικές μας, τους δικούς μας τόπους παραγωγής για να διαφυλάξουμε τις θέσεις εργασίας, για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Το energy mix, το ενεργειακό μείγμα των άλλων κρατών, βεβαίως θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη, χωρίς να προσπαθούμε απαραίτητα να αντιμαχόμαστε τα κράτη αυτά, αλλά να προχωρούμε μαζί τους για να είμαστε όλοι κερδισμένοι. Και αυτό ισχύει όχι μόνο για το ενεργειακό μείγμα, αλλά και για το περιβάλλον και για την προστασία των θέσεων εργασίας και για τις κοινωνικές προδιαγραφές. Η Ευρώπη μπορεί πάντα να είναι λίγο πιο ακριβή, ίσως λίγο πιο καινούρια ιδέα να προσφέρει, λίγο πιο καινοτόμα προϊόντα να έχει να δώσει. Και αν είναι πιο ακριβή η καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες, η δυνατότητα τη κατάρτισης και της περαιτέρω μάθηση θα είναι τα πλεονεκτήματα πάνω στα οποία μπορούμε να στηριχθούμε. Και όχι τα μειονεκτήματα που θα αποκλείουν του δικού μα ανθρώπου από τι θέσει εργασία σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Έττιγκερ, έχετε απαντήσει εν μέρος αυτό το οποίο ήθελα να σας ρωτήσω, απαντώντας για τους ε, αγωγούς αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα όμως να έχω κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες σε σχέση με τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θέλετε να ε, εγκρίνετε για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη επαρκούς διασύνδεσης στον τομέα του φυσικού αερίου μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Έτιγκερ. Μεταξύ των ε, ε, εθνικών αρχών και των περιφερειακών αρχών, οι συμφωνίες που έχουν γίνει θα πρέπει να διατηρηθούν. Αυτό αφορά και το φυσικό αέριο και όλες τις άλλες ενεργειακές πηγές. Εγώ συμφωνώ σε ό,τι αφορά το γενικότερο θέμα της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς και όχι μονάχα σε επίπεδο εθνικής, ε, εθνικών αγορών. Είναι απαραίτητο να υπάρξει πλήρη συμμετοχή των φορέων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και να αλλάξουν οι τωρινές συνθήκες. Είτε γίνεται αυτό μέσω από νέες ρυθμίσεις είτε μέσα από νέα κίνητρα οικονομικού χαρακτήρα αλλά από το παράδειγμα της δικής μου περιοχής της Βάδης Βιρτεμβέργης. Ξέρω ότι έναντι της Γαλλίας δεν υπάρχει σχεδόν καμία δυνατότητα μεταφοράς ε, φυσικού αερίου και ενέργειας και φανταστείτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο πόσο πιο δύσκολα είναι τα πράγματα. Συμπληρωματικό ερώτημα. Ευχαριστώ κύριε Έτιγκερ. Εγώ σας εύχομαι μεγάλη επιτυχία στο στόχο να μπορέσετε με μεγάλη ενεργητικότητα να αντιμετωπίσετε το, ε, το θέμα της ενέργειας. Ευχαριστώ. Το επόμενο ερώτημα, η κυρία Κορόνσκα Μπομπίνσκα. Ε, mm. Ευχαριστώ πολύ. Αναφέρατε στην εισαγωγική σας ομιλία ότι τώρα ανοίγει μια νέα περίοδος όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική. Άρα έχετε την τύχη να είσαστε ένας ιστορικός επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που διαμορφώνει και επηρεάζει αυτή την ενεργό ευρωπαϊκή πολιτική. Και σχετικά με αυτό καλοδεχούμενα αυτά που είπατε για μεγαλύτερη αλληλεγγύη και εξευρωπαϊσμό της ενεργειακής πολιτικής. Σχετικά με αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Τώρα τα κράτη-μέλη μπορεί να είναι απομονωμένα από βασικές ενεργειακές πηγές. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα εφαρμόζατε ούτως ώστε να εξασφαλίσετε την εφαρμογή της αρχής της αλληλεγγύης, άρθρο 194 της Συνθήκης της Λισαβόνας. Τι θα κάνετε για να προωθήσετε την ανάπτυξη και χρηματοδότηση της ε, νοτίας διόδου για την διέλευση φυσικού αερίου και άλλων πηγών παροχής φυσικού αερίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Για το δεύτερο ερώτημά σας. Στην ε, Νότια Ευρώπη, στην Νότια Λύση όπως λέγεται, βλέπω τη δυνατότητα να υπάρξει ένας νέος χώρος παροχής ε, φυσικού αερίου από το Αζερβαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν και βλέπω επίσης την δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε και να μειώσουμε την εξάρτηση από την Ρωσία στον τομέα του φυσικού αερίου χωρίς να διαλύσουμε την εταιρική σχέση που έχουμε δημιουργήσει με την Ρωσία η οποία θα εξακολουθήσει και στην επόμενη δεκαετία να είναι πάρα πολύ σημαντική. Και επίσης το North Stream, ο διάβλος Βαλτικής που βρίσκεται στο προήμιο της ε, υλοποίησή του θα πρέπει να είναι γεγονός ότι μία υλοποίησή του μόνο με τη συμμετοχή των βαλτικών χωρών και της με την ε, Πολωνία και τις βαλτικές χώρες μονάχα αυτό δεν θα ήταν δείγμα αλληλεγγύης. Για μένα δεν μπορούν οι διμερείς συμφωνίες μακροπρόθεσμα να εξακολουθήσουν να ισχύουν θα πρέπει να αντικατασταθούν εν καιρό από ευρωπαϊκές, ευρωπαϊκού χαρακτήρα συμφωνίες. Είμαι ε, πεπισμένος ότι ό,τι πρόκειται για μεταφορά ενεργειακών πηγών από τρίτες χώρες παραγωγής θα πρέπει οι συμφωνίες αυτές να καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά και όχι από τρίτες χώρες. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε και από τις ε, τρίτες χώρες οι οποίες είναι παραγωγή ότι δεν θα ε, θέτουν σε μειονεκτική θέση την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα δίνουν τα προϊόντα αυτά σε υψηλό επίπεδο ποιότητος και σε ανταγωνιστικές τιμές. Κύριε Κολάσκα Μπομπίσκα, θέλετε να θέσετε συμπληρωματικό ερώτημα. Ναι, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η δήλωσή σας για την Πολωνία και τις άλλες χώρες της περιοχής. Έχω λοιπόν το συμπληρωματικό ερώτημα η συμφωνία του για τον αγωγό Ναμπούκο. Εκεί συμπεραφάνονται ρήτρε διαφύλαξη για παροχή φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη-μέλη, καθώ και ε, για συμμετέχοντες στην ενεργειακή κοινότητα. Θα υποστηρίζετε παρόμοιε ρήτρε διαφύλαξη για όλα τα κράτη-μέλη, να συμπεριλαμβάνονται όλα τα κράτη-μέλη σε, άλλε σχεδιαζόμενε συμφωνίε συμφωνίες για αγωγού που μεταφέρουν ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφέρατε το Nord Stream θα συμπεριλαμβάνεται τέτοιου είδους ρήτες διαφύλαξης και στο Nord Stream και η συμφωνία Ναμπούκο θα έπρεπε να επεκταθεί και για το Ατζερμπαϊτζάν και τη Γεωργία. Τι πιστεύετε. Κύριε Ότιγκερ. Υπάρχουν υφιστάμενες συνθήκες, συμβάσεις που πρέπει να τηρηθούν, συμβάσεις με τους επενδυτές, τους προμηθευτές και βεβαίως θα πρέπει αυτές οι σχέσεις εξωτερικές να αναπτυχθούν κατά τρόπον ώστε ούτε κανείς να έχει προνομιακή μεταχείριση, ούτε κανείς να βρίσκεται σε δυσμενή θέση και ο στόχος να είναι εν τέλει η πρώτη ύλη να φτάνει σε εμάς με συνθήκες τίμιες, με ασφάλεια και προγραμματισμό να φτάνει λοιπόν μέχρι την Ευρώπη και από εκεί πέρα ο κάθε ένας ή κάθε μία μέσα στην εθνική αγορά, σε κάθε τομέα ε, της βιομηχανικής δραστηριότητας, να είναι σε θέση να αξιοποιήσει με τους ίδιους όρους αυτή την πρώτη ύλη μέσα σε μια ανοιχτή και διαφανή αγορά. Εδώ υπάρχει αρκετή δουλειά να γίνει. Για το Δένα Μπούκο, ασφαλώς θα μας πρέπει να μας απασχολήσει κατά προτεραιότητα στην εξωτερική πολιτική η ε, ερώτηση του πώς μεταχειριζόμαστε κράτη τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές όπως έχουν αυτές συμφωνηθεί. Από την άλλη, η ενέργεια είναι πρώτη ύλη, προϊόν. Και πρέπει να την αναζητούμε εκεί που προκύπτει, εκεί που παράγεται και να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες μας για συμπληρωματικές προελεύσεις ενέργειας. Εδώ έχει ένα ρόλο να δραματίσει το Αζερβαϊτζάν. και θα πρέπει να εξετάσουμε και για εφέτος εάν υπάρχει δυνατότητα να συνεχιστεί η προμήθεια, εάν πρόκειται να κλείσει, εάν θα προχωρήσει περαιτέρω τον Αμπούκο. Αυτό θα αποφασιστεί εφέτος. Παρακαλώ. Η επόμενη ερώτηση. Redan framkommit finns det Κύριε Έτιγκερ, όπως ελέγχθη ήδη, υπάρχει η ανησυχία ότι είσαστε πολύ κοντά σε μεγάλα βιομηχανικά συμφέροντα και ότι θα υποστηρίξετε παραδείγματος τομείς ενέργειας όπως η πυρηνική ενέργεια. Η ενέργεια. Θα θέσετε σε, σε, σε πρώτο επίπεδο τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία του περιβάλλοντος. Το 2007 ήδη είχατε συμμετάσχει σε μια δεξαμενή σκέψεως η οποία είχε συνδεθεί αυτή η δεξαμενή σκέψη με αντισημιτικές ε, εκδηλώσεις απόψεων. Θα ήθελα να ξέρω αν αυτό θεωρείται ότι είναι συμβατό με τις προτεραιότητές σας, κύριε Έτουγκερ. Καταρχάς, κύριε Βουλευτά, δεν έχω ούτε από την ε, AWE, ούτε από την ΕΟΝ, ούτε από την NDF μετοχές. Καθήκον μου όμως ήταν πάντοτε να έχω επαφές και να διατηρώ τις επαφές με τις επιχειρήσεις. Δεν είναι δυνατόν η πολιτική κατά τη δική μου έποψη να αποκοπεί από τον επιχειρηματικό κόσμο. Πρέπει να είναι σε διάλογο με τον επιχειρηματικό κόσμο. Όπως και το το η Μετάλ της Γερμανίας πρέπει να έχει επαφή με την κυβέρνηση όπως και η ΕΝΤΕΦ η οποία προσφέρει κατά 45% το, την προμήθεια ενέργειας, τους, τον εφοδισμό ενέργειας για τη Βάδη Βιρτεμβέργη, προφανώς είναι για μένα συνομιλητές, ε, μονάδες με τις οποίες θα έχω ανταλλαγή απόψεων και από τις οποίες θα αποκομίσω κάποια στοιχεία για να προχωρήσω λήψη αποφάσεων. Εδώ δεν είναι ζήτημα όμως. Δεν τίστε να αμφιβόλω η ανεξαρτησία κανενός. Γιατί τι αποφάσει για οποιοδήποτε θέμα ενέργεια στα μέχρι τώρα καθηκοντά μου πάντοτε μπόρεσα να διαφυλάξω την ανεξαρτησία μου κατά απόλυτο τρόπο. Γιατί δεν δεύτερη σα ερώτηση. Ο προκάτοχός μου ήταν ε, μέλος σε μία ένωση δραστηριοτήτων, ωστόσο εγώ μπορεί αυτόματα να κληρονόμησα αυτή τη συμμετοχή, τη διδιότητα του μέλους, χωρίς όμως ποτέ να πάω να συμμετάσχω σε συνεδριάσεις, σε ε, οργανώσεις τέτοιες. Το ίδιο είναι και το ζήτημα του αντισημιτισμού στην χώρα μου και στην ιδιαίτερη μου πατρίδα πάνω απ' όλα. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα και η σχέση μου με την ε, κοινότητα την εβραϊκή ε, είναι πάντοτε ανοιχτές, καθαρές και δεν επηρεάζουν την πολιτική μου κρίση. Πιστεύω ότι καθήκον μου είναι να επιτελέσω τα καθήκοντα τα οποία μου ανατίθενται εδώ στις Βρυξέλλες. Παρακαλώ, η συνάδελφος για συμπληρωματική ερώτηση. Ε, Ευχαριστώ για, το, για την απάντησή σας. Πώς ε, ορίζεται την έννοια της σύγκρουσης συμφέροντος μέσα στα πλαίσια του κώδικα συμπεριφοράς της ε, Κομισιόν. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μνήμα αυτής της έννοιας. Νομίζω θα ήταν σημαντικό οι τι ακριβώς σημαίνει σύγκρουση συμφερόντων για αυτούς και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας στάση σε σχέση με το θέμα αυτό για να αποφευθούν οι συγκρούσεις ε, συμφερόντων και όχι μονάχα οι επαφές με ορισμένους κύκλους. Κύριε Έτουγκερ, μιλήσα για ανεξαρτησία. Χρειάζεται δικαιοσύνη έναντι όλων αυτών με τους οποίους έχω κάποιες υποχρεώσεις λόγω του αξιώματός μου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράγραπτο μέσα σε μια δημοκρατία και ένα δημοκρατικό κράτος δικαίου. Τώρα υπάρχει ίσως κάποιο σύστημα για την αντιμετώπιση των ε, συμφερόντων των ε, επιτρόπων, το οποίο είναι το σύστημα αυτό είναι πιο ε, ισχυρό από ότι οποιοδήποτε άλλο σύστημα το οποίο ισχύει παραγματικά σε επίπεδο εθνικών κρατών και επίσης στην περίπτωση των βουλευτών. Στην περίπτωση της ε, Γερμανικής Βουλής το θέμα αυτό των λόμπι έχει αντιμετωπιστεί ενδελεχώς. Αλλά η Κομισιόν ελέγχεται πολύ περισσότερο από ότι οποιοδήποτε άλλος. Νομίζω λοιπόν ότι πέραν όλων των ε, προδιαγραφών αυτό το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι η πρακτική συμπεριφορά του κάθε επιτρόπου και ο τρόπος με τον οποίο καθορίζει ο καθένας την ανεξαρτησία του και τα καθήκοντά του. Και εγώ βασίζομαι στην αρχή της ανεξαρτησίας και της επιζήτησης της ισοδικίας έναντι όλων αυτών με τους οποίους εγώ έρχομαι σε επαφή. Και σε ό,τι αφορά την επιρροή των λόμπι, των ιδιαίτερων συμφερόντων, των ε, όλων αυτών των ε, θεμάτων, εγώ δεν θα επηρεαστώ, είναι το δικαίωμά τους να ασκήσουν την, άποψη, την ε, δράση τους και είναι δικαίωμα όλων να ελέγχουν το άτομό μου ακόμα και με επιβητικό τρόπο. Κυρία Σίζελη. Ευχαριστώ κύριε Έτιγκερ. Στην εισαγωγική σας δήλωση είπατε ότι ένας από τους πυλώνες της ενεργειακής πολιτικής ήταν και η βιωσιμότητα και τονίσατε την ενεργειακή απόδοση χαμηλές εκπομπές άνθρακος και οι πηγές που εκπέμπουν χαμηλά επίπεδα άνθρακο είναι σημαντικέ συμπεριλαμβανομένε πυρηνική ενέργεια. Όλα αυτά απαιτούν μεγάλε επενδύσει, τεράστιε επενδύσει. Πολλά κράτη-μέλη ανακοίνωσαν επέκταση των πυρηνικών του προγραμμάτων και θα ήθελα να ξέρω πώ πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει να διαμορφωθεί ένα σταθερό ε, περιβάλλον για τέτοιου είδου επενδύσει. Και κάτι άλλο. Φέτο περιμένουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει πρόταση οδηγίας όσον αφορά τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων. Ποιο θα πρέπει να είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτω ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή αποκομιδή των ραδιενεργών καταλήπων και πώ θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά αυτή την ασφαλή μεταφορά αυτών των αποβλήτων. Κύριε Σέτσιγκερ. Έχουμε να κάνουμε με επενδύσεις που αφορούν συνολικά τις ενεργειακές μας υποδομές. Αυτό θα πρέπει να είναι ο στόχος μας, γιατί μόνο με αυτές τις επενδύσεις μπορούμε να μειώσουμε τις εξαρτήσεις μας και να αναπτύξουμε μακροπρόθεσμες οικολογικές προοπτικές. Και έτσι θα πρέπει την επόμενη χρονιά να εξετάσουμε ποια είναι η κατάσταση στον κόσμο μας, ποια είναι η διαμόρφωση περιβαλλοντική, τι κάνουμε στην οικονομία, τι κάνει ο πολίτης, τι είδους τέλη, φόροι, προγράμματα αναπτύσσονται, τι είδου συνεργασία μπορούμε να έχουμε με ευρωπαϊκές τράπεζες και σχετικά προγράμματα δανειοδότησης για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών, με ένα πεδίο κινήτρων, κατά την άποψή μου, με δυνατότητες που μπορεί να μας προσφέρει ο προϋπολογισμός, διότι μέχρι τώρα είχαμε πολλά μεμονωμένα μέτρα, μια πληθώρα μεμονωμένων μέτρων, αλλά όχι μια ενιαία και οργανωμένη προγραμματισμένη πολιτική. Πρώτον. Και δεύτερον, όσον αφορά την αποκοδημίδη και τα φύ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, αυτό μπορεί κανείς, αυτό πρέπει κανείς, είτε είναι υπέρ είτε είναι κατά της πυρηνικής ενέργειας, να το αντιμετωπίσει με σοβαρότητα. Είναι μια δύσκολη περίπτωση, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Έχουμε πολλά απόβλητα, ειδικά απόβλητα όπως λέγονται, είτε πυρηνικά είτε άλλου είδους ε, τοξικά απόβλητα. Και πρέπει ε, να δούμε ότι οργανώσαμε τον τρόπο αυτό αποκοδμιδίσει τα ε, σε μια εποχή που ήταν ευνοϊκή για την ανάπτυξη των χώρων ή των επιλογών των γεωγραφικών. Αυτά ανεξαρτήτως των επιλογών για το μέλλον της πυρηνικής παραγωγής, πυρηνικής ενέργειας. Πρέπει και χωρίς ε, μόνο να περιοριζόμαστε στον ε, γνώμονα του κόστους, να εξετάσουμε πλέον γενικά, ε, συνολικά, το θέμα της αντιμετώπισης αυτών των αποβλήτων. Πιστεύω, πιστεύετε μάλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα επίπεδο, ένα πλαίσιο προδιαγραφών για την αποκομιδή των πυρηνικών αποβλήτων και για την κατάργηση λειτουργίας εγκαταστάσεων που θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να χρηματοδοτείται ανεξάρτητα. Κύριε Σότνικερ, φαντάζομαι ότι προβλέπω δηλαδή ότι η ευρωπαϊκή ε, διάσταση και για την έρευνα αλλά και για την διαβούλευση θα πρέπει να αναλάβει ε, δραστηριότητα και επιπλέον θα πρέπει να προσδιορίσει πιστεύω και τις προδιαγραφές. Προδιαγραφές ασφαλείας, προδιαγραφές οικολογικές, καθήκοντα συγκεκριμένους στόχους δηλαδή τους οποίους θα πρέπει να επιτελέσουν είτε οι επιχειρηματίες, είτε οι επενδυτές, είτε οι κυβερνήσεις, το κράτος, έτσι ώστε να μην ε, προκύψουν στην υπόθεση αυτή ε, διαφορές που θα επηρέαζαν είτε την αηφορία είτε την ασφάλειά μας στην υπόθεση αυτή. Ευχαριστώ κύριο Σφόποντα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Έτιγκερ, αν μπορώ να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα μετά από αυτό το οποίο απαντήσατε. Μιλήσατε για τα υψηλά επίπεδα ασφαλείας, για την πυρηνική ενέργεια. Πιστεύω και εγώ ότι θα πρέπει να δώσουμε να, αν θα πρέπει να δώσουμε το υψηλότερο δυνατό επίπεδο σε τεχνικό, από τεχνική άποψη ή ένα χαμηλότερο. Και χαιρετίζω αυτό το οποίο είπατε ότι δεν πρέπει να γίνονται πια διμερείς συμβάσεις σε ό,τι αφορά την ε, προμήθεια ενέργειας. Πώς θα το επιτυχετε αυτό, θα ζητήσετε από το Κοινοβούλιο να απαγορευτούν αυτές οι, οι διαδικασίε διμερών συμφωνιών ή να υπάρχει προηγουμένω μια ακρόαση, μια συμφωνία με την Κομισιόν, να έχει τη δυνατότητα η Κομισιόν να θέτει ενστάσει. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή η βασική αρχή την οποία εγώ χαιρετίζω, πώ ακριβώ θα την εφαρμόσετε στην πράξη. Κυρία Τουγκέ, παρακαλώ. Κύριε Σφόμποντα. Το άρθρο 194 αναφέρεται στην αλληλεγγύη. Το πνεύμα της αλληλεγγύης θα πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη και για την αγορά ενέργειας και θα πρέπει να δεσμεύει όλους. Αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορούν τα νέα κρατημέλη να ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά αυτές τις συμβάσεις. Αυτό σημαίνει ότι όταν έρχεται ένα αγωγός όπως ο Ναμπούκο παραγωγικά από την Τουρκία ω την Αυστρία θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα όλες οι χώρες να ευνοούνται και καμία να μην βρίσκεται σε μειονεκτική θέση. Σε ό,τι αφορά τις, ε, τα οικονομικά συμφέροντα είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην λήψη συγκεκριμένων μέτρων τα οποία θα εξασφαλίσουν την εφαρμογή της αλληλεγγύης να μην υπάρξει μειονεκτική μεταχείριση ορισμένων κρατών και να υπάρξει η ίδια ασφάλεια σε ό,τι αφορά όλες τις χώρες μας σε νομικό επίπεδο. Είμαι απόλυτα έτοιμος λοιπόν να προχωρήσουμε αποφασιστικά με τη βοήθειά σα και να θεσπίσουμε νομικά δεσμευτικέ ρήτρε για τα ζητήματα αυτά. Κύριε Σφόποντα, για συμπληρωματικό ερώτημα. Νομίζω ότι είναι καλή η απάντησή σα, κύριε Έτιγκερ. Ελπίζω ότι δεν θα είστε μονάχα διαθέσιμος να κάνετε αυτές τις πρωτοβουλίες, αλλά ότι θα καρποφορήσουν αυτές, γιατί είναι απαραίτητο αυτό το κοινό συμφέρον μας να γίνει πραγματικότητα. Τώρα, για το θέμα της ε, Υψηλή ασφάλεια στην πυρηνική ασφάλεια. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο ασαφές. Είναι αυτό το οποίο είναι ε, το τεχνικά επιτευκταίο ή αυτό το οποίο εσείς θα θεωρήσετε σε μια συγκεκριμένη στιγμή επαρκές. Εμείς μιλάμε για τις νέες δυνατότητες οι οποίες δημιουργούνται. Επομένως, το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που είναι εφικτό, χωρίς να δημιουργήσει υπέρογκο κόστος και άλλους περιορισμούς που δεν μπορεί η οικονομία μας να τους αντέξει. Κύριος Εδώ είμαι στα δεξιά. Κύριε Έτικερ, μία από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι ανοιχτή και λειτουργική εσωτερική αγορά στον τομέα της ενέργειας Όλοι θέλουμε να υπάρχει ασφαλής ενεργειακός εφοδιασμός. Και ένας από τους σημαντικούς τρόπους για την βελτίωση της καταστάσεως είναι μέσω της χρήσεως ανοιχτής λειτουργικής ενεργειακής αγοράς. Δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ενεργειακές νησίδες απομονωμένες από τη, τα κοινά ενεργειακά δίκτυα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι οι βαλτικές χώρες, που είναι 100% απομονωμένες αφορά το φυσικό αέριο και σχεδόν πλήρω απομονωμένε χώρε από το κοινό ενεργειακό δίκτυο. Το ερώτημά μου είναι απλούστατο. Τι θα κάνετε ως Επίτροπος για να αποφύγετε την απομόνωση κάποιων κρατών μελών όσον αφορά το ενεργειακό δίκτυο και να αυξήσετε ε, τον ασφαλή εφοδιασμό, τον ενεργειακό. Κύριε Έτσιγκερ, έχετε το λόγο. Η γεωγραφική κατάσταση αλλά και η κατάσταση των υποδομών στις ε, βαλκανικές χώρες στις βαλκανικές χώρες είναι γνωστή σε μένα, είμαι εξοικειωμένος με αυτή και δεν πρέπει βέβαια να παραμείνει έτσι, πρέπει να βελτιωθεί, πρέπει να αναπτυχθούν τα δίκτυα, οι υποδομές και για το φυσικό αέριο και για τον ε, ηλεκτρισμό. Και θα ήθελα να σημειώσω ότι τα μεγάλα ευρωπαϊκά δίκτυα ή καλύτερα διευρωπαϊκά διυπηρωτικά δίκτυα δεν μπορεί ίσως να φτάσουν σε όλα τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα και στον ίδιο βαθμό, αλλά πάντως θα πρέπει να υπάρχει το επαρκές περιεχόμενο για την περαιτέρω διαβίβαση στο πλαίσιο ενός ε, εσωτερικού ευρωπαϊκού δικτύου, έτσι στο καθένας να έχει την κατάλληλη τεχνολογική ε, υποδομή και οικονομική ε, δυνατότητα ώστε να αξιοποιήσει αυτές τις δυνατότητες και να ικανοποιήσει τις ανάγκες του. Πρέπει λοιπόν να απτύξουμε ε, προγράμματα δικτύων για τα επόμενα χρόνια που σημαίνουν ταυτόχρονα ανάπτυξη δυνατοτήτων, δηλαδή μείωση των εξαρτήσεών μας. Αυτό όμως το να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τα έξω δεν σημαίνει ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ε, εξάρτησή μας προς τα έσω, προς άλλα κράτη. Κύριε Κάρεν, συμπληρωματική. Σας ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να ενισχύσει την επιρροή της αναφορά της αποφάσεις συγκεκριμένων κρατών μελών όσον αφορά τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές όταν αυτές οι αποφάσεις ίσως να οδηγούν σε απομόνωση άλλων κρατών μελών. Ευχαριστώ. Οι επενδύσεις θα πρέπει να στοχεύουν περισσότερο τους φορείς εκείνους που είναι οι ιδιοκτήτες, οι επιχειρήσεις διανομής για την ποιότητα, τον εξυγχρονισμό και την αποτελεσματικότητα των δικτύων μας. Έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ο κύριος Χατζημακάκης έχει το λόγο. Με μια παράκληση, κύριε Τσιγκέρ. Αν θέλετε να στρέφεστε περισσότερο προς το μικρόφωνο, διότι δυσκολεύεται πολύ το έργο των διερμηνέων. Κύριος Χατζημαρκάκης. Πρόεδρε, Κύριε Έτσιγκερ, βλέπω ότι είσαστε γερός, ε, γερά κατσμένος στον ε, θόκο σας και χαίρομαι ιδιαίτερος. Ναι, βλέπω ότι θα μου κόψετε χρονομιλίας όμως, Πρόεδρε. Αλλά μας μιλάτε για τον Baden-Württemberg ε, και πώς λειτουργεί και όλα αυτά. Τα ξέρετε πολύ καλά και μπράβο σας. Πλην όμως, οι κατευθυντήριε γραμμέ, τι οποίε έχει συμπεριλάβει στην ενημερωτική του επιστολή προ εσά και εμά, βέβαια, ο κύριο Μπαρόσο βλέπω ότι δεν έχουν τόσο πολύ τη προσοχή σα. δεν τι έχετε τόσο πολύ αναπτύξει. Εμένα με ενδιαφέρει το, η ευρωπαϊκή διάσταση, τα ευρωπαϊκά οράματα και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και συγκεκριμένα πώ θα χειριστείτε τα κράτη-μέλη. Εσεί ο ίδιο είπατε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διαθέσουν περισσότερα χρήματα, ότι θα πρέπει να προχωρήσουν στην εφαρμογή περισσότερων ε, προγραμμάτων για την ε, ηλιακή τεχνολογία. Οι σε παραδείγματι, έχουν την πιο σύγχρονη τεχνολογία ε, νομοθεσία συγγνώμη, του κόσμου για την ηλιακή ενέργεια, αλλά δεν την εφαρμόζουν. Τι θα κάνετε λοιπόν για αυτά τα πράγματα, τι θα κάνετε, είστε διατεθειμένο να ανεβείτε στην αρένα και να πυγμαχίσετε με του ε, ε, άλλου επιτρόπου, αλλά πάνω απ' όλα με του πρωθυπουργού και του καγκελάριου. Κύριε Έτιγκερ, είδατε, είδατε ότι ήρθε η ώρα των αθλητικών ε, ειδήσεων. Παρακαλώ. Κύριε Έτιγκερ, εχθές ακόμη μου συνέστησαν διάφοροι συνάδελφοι από διάφορες πλευρές θα πρέπει να πω ότι θα πρέπει να αποφύγω τις κατευθυντήριες γραμμές ε, και να ε, μείνω πιο περιορισμένο στις δηλώσεις μου. Ναι, θα πρέπει να πω ότι οι κατευθυντήριες γραμμές ισχύουν, είναι συλλογικό όργανο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είμαστε υποχρεωμένοι να συμβαστούμε τις κατευθυντήριες γραμμές. Πλην όμως θα πρέπει και να τις ε, διευρύνουμε τα επόμενα 4-5 χρόνια, να τις εφαρμόσουμε και να τις διευρύνουμε. Και βέβαια έχω και εγώ τις δικές μου ιδέες να προσφέρω σε αυτήν την υπόθεση. Γιατί να σας πω το εξή. Έδειξε ένα πράγμα η Κοπεχάγη, ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, λειτουργεί στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή, τότε χάνει ολόκληρο ο κόσμο. Δεν πρόκειται για την Κίνα, δεν πρόκειται για τον έλεγχο των μέσων μαζική ενημέρωση, δεν πρόκειται για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Μόνο με σαφείς ε, επιλογές, μόνο με αλληλεγγύη και κοινή δράση μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τώρα ειδικά, μέσα στην κρίση, αλλά και μετά την κρίση, εγώ είμαι διατεθειμένο αυτό να τηρήσω. Αυτό ισχύει τώρα με την Κοπεχάγη, αυτό ισχύει τώρα με τη συνθήκη. Η ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει διαρκώ να διονγκώνεται, να επεκτείνεται και θα πρέπει κάθε δυνατότητα που μα προσφέρεται να την αξιοποιήσουμε. Καθήκον μα κοινό μας καθήκον είναι όχι μόνο την αποδοχή σε όλη την Ευρώπη και την ορατότητα της Ευρώπης για τον πολίτη να ενισχύσουμε, αλλά ταυτόχρονα και να συμβάλλουμε στο ότι τα επόμενα χρόνια η, ε, Ευρω... η ζωή μας η νομοθεσία μας, οι δράσεις μας θα αναπτυχθούν κατά τρόπο ευρωπαϊκό, εξευρωπαϊσμένο, όχι δηλαδή με την έννοια της κεντρικής οργάνωσης και διοίκησης από ένα μόνο κέντρο, αλλά της κοινοτικής κοινή προσπάθεια. Έτσι τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Ο κύριο Χατσιμαρκάκη έχει συμπληρωματική ερώτηση. Πολύ συγκεκριμένα να επιμείνω με ένα μου παράδειγμα για να δούμε σε ποιο βαθμό είστε σε θέση να επιβάλλετε συγκεκριμένε προδιαγραφέ, παγκόσμιε προδιαγραφέ, όπω άλλωστε είχε κάνει και ο προκάτοχό σα σε ένα βαθμό, αλλά και πόσο μπορείτε με του ε, με τους ε, λοιπού επιτρόπου, τον κύριο Ποτόσνη και ιδιαίτερο, αλλά και του έξω εταίρου ε, Κίνα και λοιπού να ε, βρείτε λύσεις. Εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαρκώς επιμένουμε για την παραγωγή ε, είτε στις οικιακές συσκευές, είτε στα ηλεκτρονικά, ε, στα θέματα προστασίας του καταναλωτή. Όμως τον έχουμε να κάνουμε με μεγάλες τουρμπίνες, με, μεγάλη, με βαριά βιομηχανία. Μπορείτε εσείς ε, σε σχέση με τη Βάδη τη παραδείγματι, να κάνετε κινήσεις αντίστοιχες για την Ευρώπη και να, να, αγωνιστείτε για τα συμφέροντα της Ευρώπης όπως αγωνιστήκατε για τα συμφέροντα της Βιτεμβέργης. Ο πρόεδρος, ναι, αλλά ένα λεπτό, μην απαντήσετε για τη Βάδη αλλά για την Ευρώπη. Απάντησε ο κ. Σέτιγκερ. Ναι, και άλλωστε το έχω κάνει. Και όταν έχουμε να με μακροπρόθεσμο η ασφάλεια των, ε, του προγραμματισμού, μπορούμε εμείς η Ευρώπη να αποτελέσουμε στοιχείο ωφέλους, κέρδους για τις επιχειρήσεις μας. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη έρευνα για την ενέργεια. Μπορούμε χάρη στα δίκτυα των ε, εθνικών ερευνητικών κέντρων γιατί ήδη τώρα έχουμε ξεκινήσει με μια πρώτη προσπάθεια ίδρυση στατιών ερευνητικών κέντρων και με τα καθήκοντα που θα προσδιορίσουμε μπορούμε να επιτρέψουμε στη βιομηχανία να γνωρίζει τι έχει να επιτελέσει, προς τα που πηγαίνει και ταυτόχρονα να προαγάγουμε τις προδιαγραφές που ισχύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ως εκ τούτου, εγώ και στον τομέα της βιομηχανίας, στον βιομηχανικό κλάδο και όχι μόνο στην ε, βιομηχανία, στον κλάδο μάλλον παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά γενικότερα στην βιομηχανική παραγωγή, εγώ προσωπικώς είμαι διατεθειμένος να εμπλακώ ενεργά για να υποστηρίξω την ανάπτυξη του δυναμικού που υπάρχει, γιατί ξέρω ότι υπάρχει και για ανανεώσιμες πηγές και για αποτελεσματικότητα και για ε, καλύτερα και οικολογικά κτίρια, γιατί υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Γιατί για τις μικρές συσκευές, θα είναι οικιακές, θα είναι ε, τα hi-fi, είτε είναι ηλεκτρονικές άλλες συσκευές. Πολλά έχουμε κάνει, αλλά στις, ε, στις, ε, στη βαριά βιομηχανία έχουμε ακόμη πολλή δουλειά. Παρακαλώ, επόμενη ερώτηση. Κύριε Σότσεφ, ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς, να συγχαρώ τον κύριο Έτιγκερ για το διορισμό του. Ενεργειακή απόδοση είναι το θέμα του ερωτήματός μου. Τι δυνατότητες υπάρχουν για να δημιουργηθεί μια οικονομία με χαμηλέ εκπομπές ε, ενέργειας. Είναι κάτι που τονίζεται ότι είναι σημαντικό. Το σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα είναι πολύ σημαντικό εργαλείο στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη του στόχου του 20%. Μπορείτε παρακαλώ να περιγράψετε τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου αυτού σχεδίου δράσεως, το επικείμενο σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Και ανάλογα με τις απαντήσεις σας, μάλλον βλέπω ότι χρειάζονται περισσότερες ε, επενδύσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα. Γι' αυτό το νέο σχέδιο δράσης θα οδηγούσε σε κάποιες οικονομικές απαιτήσεις για ενεργειακή αποδοτικότητα έχω υπόψη μου το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο τόσο ώστε να μπορεί να χρηματοδοτηθεί αυτή η δημιουργία της βάσος για μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Κύριε η αποδοτικότητα ενέργειας για τα ιδιωτικά κτίρια είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Και έχουμε ξεκινήσει προγράμματα εξυγίανσης για τα κτίρια και είχαμε θετικές εμπειρίες με αυτά τα προγράμματα. Θα ήθελα λοιπόν να έχω προγράμματα τα οποία θα δώσουν κίνητρα σε συμφωνία με εθνικές και περιφερειακές αρχές να τα αναπτύξουμε περισσότερο. Όχι μόνο θα προωθήσουν την ποιότητα ζωής στη στέγαση και την ε, ομορφιά των κτίριων κατά κάποιο τρόπο, αλλά συγχρόνως θα εξασφαλίσουν ότι τα κτίρια αυτά έχουν καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά και θα βελτιώσουν την ε, κατάστασή τους από αυτή την άποψη. Αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται στην ε, διαδικασία των, ε, της παραγωγής ενέργειας. Τα κτίρια λοιπόν παραγωγής, ε, τα γραφεία, όλα τα κτίρια θα πρέπει <clears throat> να ακολουθήσουν αυτή την οδό και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια εν γέννη και να χρησιμοποιήσουμε ως το δυνατόν τις καλύτερες μεθόδους. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τον παράγοντα της εκπομπής διοξιδίου του άνθρακος για τις μεταφορές. Για μένα όμως η δυνατότητα μεταφοράς του ηλεκτρισμού με χαμηλές απώλειες είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να διαδραματίσει και στην έρευνα και στην παραγωγή ε, οχημάτων Όσο αφορά επίσης και τη δημιουργία ευφυών δικτύων, θα πρέπει να εξυπηρετήσει την εσωτερική κινητικότητα. Κανένας άλλος από, σε όλο τον κόσμο δεν έχει τόσο σημαντικές προκλήσεις όσο εμείς και εμείς πρέπει να γίνουμε το κέντρο της καινοτομία για τα θέματα αυτά. Κύριε Ούτσερ. Ε, Η συμπροματική μου ερώτηση για να πετύχουμε 20% μείωση της κατανόλωσης πρωτογενούς ενέργειας, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στη βιομηχανία για να επενδύσει. Απ' την άλλη πλευρά, αυτή στο νέο σύστημα ε, ανταλλαγής ρήπων, εμπορίου ρήπων, επιβάλλουμε ένα φόρο στη βιομηχανία μας με το προτινόμενο σύστημα δημοπρασιών και μειώνουμε τη δυνατότητα για επενδύσεις. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό. Θεωρώ ότι τα εργαλεία της αγοράς, όπως παραδείγματος χάρη οι αδειοδοτήσεις και η εμπορία των ε, εκπομπών είναι σημαντικά εργαλεία. Δεν θέλω να αποκλείσω φορολογικά μέτρα, αλλά όταν πρόκειται για φορολογικά μέτρα, ξέρετε ότι οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ιδιαίτερα περιορισμένες. Χρειάζεται να τηρηθεί η αρχή της ομοφυγωνία και φυσικά υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις από την πλευρά των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Η εισαγωγή νέων φόρων δεν μου φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Επόμενο ερώτημα. Η κυρία Ποδηματά. Είναι πίσω σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε με κύριε Προτινόμενο Επίτροπε να σας καλωσορίσω κι εγώ από την πλευρά μου. Θα επανέλθω σε ένα θέμα που συζητήθηκε αρκετά και που περιλαμβάνεται και στις γραπτές απαντήσεις που μας δώσατε στο θέμα της πυρηνικής ενέργειας. Λέτε λοιπόν στις γραπτές απαντήσεις που μας προωθήσατε ότι θα προωθήσετε την ασφαλή χρήση της πυρηνικής ενέργειας και παράλληλα βεβαίως διευκρινίζετε ότι δεν θα φυγεί η διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να επιλέγουν το ενεργειακό τους δείγμα. Επειδή θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτή η απάντηση επιδέχεται πολλαπλών ερμηνεών και επειδή μιλήσαμε πριν και ορθώς με βάση και τη συνθήκη της Λισαβόνας για την ευρωπαϊκοποίηση της ενεργειακής πολιτικής, ήθελα να σας ρωτήσω ευθέως εάν πιστεύετε ότι η πυρηνική ενέργεια θα πρέπει να ενταχθεί σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκοποίηση της ενεργειακής πολιτικής ή αν θα πρέπει να μείνει εκτός αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ήταν η πολιτική που ακολουθήθηκε τα προηγούμενα χρόνια και εφαρμόστηκε και από τον προκάτοχό σας Επίτροπο κύριε Έτιγκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε μια νέα, μια νέα συνθήκη η οποία έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόσφατα και θα πρέπει να είναι το η βάση της εργασίας μας, η συνθήκη της Λισαβόνας. Και η συνθήκη της Λισαβόνας αναφέρει ότι η απόφαση της ε, συγκεκριμένης εφαρμογής του ενεργειακού μείγματος βρίσκεται απόλυτα στα χέρια των κρατών μελών. Το θέμα του 20% είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ένα 20% ανανεώσιμε ενέργεια σημαίνει κατά μέγιστο όρο 80% ορυκτά καύσιμα. Και είναι γεγονός ότι μπορεί κανείς να έχει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους θα καλύψει αυτό το ποσοστό με άλλους τρόπους. Μπορεί να έχουμε λοιπόν αυτό το στόχο του 20% αλλά μετά πρέπει να σκεφτούμε και για τους στόχους για τα επόμενα χρόνια, τα 50%. Το 2050 παραδείγματος Νομίζω ότι οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν στο επίπεδο στο οποίο βρίσκονται σήμερα. Υπάρχουν χώρες παραδείγματος που δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν την πυρηνική ενέργεια, Όπω η Αυστρία. Ενώ υπάρχουν άλλε χώρε όπω η Γαλλία που είναι έτοιμε να προχωρήσουν στην κατασκευή περαιτέρω πυρηνικών ε, εργοστασίων. Και στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως σας είπα προηγουμένω, βλέπω από τη μία μεριά ανάπτυξη αιωλικών πάρκων υπερακτήρων και από την άλλη μεριά προώθηση τη πυρηνικη ενεργεια επομενω η κάθε κυβέρνηση έχει μία άποψη η οποία δεν πρέπει να περιοριστεί από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ λοιπόν ως δημοκράτης δεν μπορώ να παραγνωρίσω την πολυμορφία που υπάρχει μέσα στην Ευρώπη και επομένως το δικό μας καθήκον θα πρέπει καταρχήν να είναι να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν οι προδιαγραφές ασφάλειας, ότι υπάρχει δυνατότητα να προμηθευόμαστε βασικές πηγές ενέργειας όπως το ουράνιο χωρίς κίνδυνο ασφάλειας σε διεθνές επίπεδο, να προωθήσουμε το έργο της, Ευρω... της Ευρατόμ και από εκεί πέρα το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να πάρει τις δικές του αποφάσεις. Αυτό είναι ένα δημοκρατικό θέμα. Εγώ δεν είμαι ο υπέρμαχος της πυρηνικής ενέργειας. Νομίζω απλώς ότι μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής λειτουργεί αρκετά καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Ποδηματά. Θεωρώ πολύ σαφή την απάντησή σας και την εκλαμβάνω και ως ε, δέσμευση για τη θητεία σας. Θα ήθελα λοιπόν να δω μήπως μπορούμε να αποσπάσουμε μία ακόμα δέσμευση από την πλευρά σας που αφορά στην... Είναι εντάξει με... Έχουμε... Οκ. Okay. Okay. It's okay. It's okay. Okay. Θα ήθελα λοιπόν να δω αν μπορούμε να αποσπάσουμε μία ακόμα δέσμευση από την πλευρά σα. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για την πρόθεση ενεργειακή αποδοτικότητα και πολύ ορθώ, γιατί είναι καθοριστικό στοιχείο για την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών όπως γνωρίζετε πολύ καλά στο πλαίσιο του κλιματικού ενεργειακού πακέτου που έχουμε υπερψηφίσει οι στόχοι της προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών είναι νομικά δεσμευτικοί. θα υποστηρίξετε να αναλάβουν τέτοιο χαρακτήρα νομικά δεσμευτικό και ο στόχος της προώθησης ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 20%. Σα Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Κυρία Τιγκέρα, έχετε το λόγο. Αναμένουμε στους επόμενους μήνες και στα επόμενα χρόνια να εξασφαλίσουμε την εφαρμογή συγκεκριμένων και δεσμευτικών στόχων και δεν θα πρέπει να αποτύχουμε στην επίτευξη των στόχων αυτών. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει κίνδυνος για αυτούς τους στόχους. Θα πρέπει αυτοί οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν προς μια κατεύθυνση να προχωρήσουν μέσα στα πλαίσια μιας εθελοντικής συμφωνίας. Όταν όμως υπάρχει κίνδυνος να αποτύχουμε στην επίτευξη των στόχων μας, θα πρέπει να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να αποσύσουμε αυτό τον κίνδυνο ο πραγματικός στόχος μας, αυτό που είναι η ουσία, είναι να επιτύχουμε πράγματι αυτούς τους στόχους. Και τα εργαλεία εξυπηρετούν τους στόχους. Η χρήση δεσμευτικών μέτρων είναι μονάχα σε επίπεδο ultima ratio. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε μονάχα αν δεν υπάρχει καμιά άλλη λύση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούτι Κόφερ. Μιλήσατε για εμπιστοσύνη με τον κύριο Τούρμες. Εγώ θα σας πω ότι σας εμπιστεύομαι όταν είσαστε σαφείς σε αυτά τα οποία λέτε. Και θέλω να θέσω ορισμένα ερωτήματα συμπληρωματικού χαρακτήρα. Αυτό το οποίο αναφέρατε προηγουμένως, απαντώντας στην κυρία Ποδηματά. Αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο του 20% και δεν τα δεν θα τα επιτύχουμε αυτό. Πότε θα αποφασιστούν τα μέτρα αυτά, τα νομικά, τα οποία θα είναι δεσμευτικά. Εάν λοιπόν χρειαστείτε να θεσπίσετε δεσμευτικά μέτρα, πότε θα μπορέσει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος. Και σας παραπέμπω σε αυτό που είπατε ότι μπορεί να είναι απαραίτητα πιο οξέα, πιο ισχυρά νομικά εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε απειλές, να μην επιτύχουμε τους στόχους στους οποίους θα έχουμε θέσει. Για παράδειγμα, η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία είχε ακολουθήσει την οδό των εθελοντικών στόχων και είπε τελικά όχι δεν θα μπορέσουμε μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα να μειώσουμε τις ε, εκπομπές καυσαερίων. Ένα δεύτερο ερώτημα μέσα στα πλαίσια των στόχων της εξωτερικής πολιτικής ενέργειας είσαστε έτοιμος να χρησιμοποιήσετε τον, την οδό των εμπορικών συμφωνιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήσεις ήταν. Ας προσπαθήσουμε. Ναι. Α, α, απερίφραστα ναι σε συνεργασία και συμφωνία με τον αρμόδιο για τα εμπορικά επίτροπο συνάδελφο. Και τα εφιστάμενα προγράμματα δράσης ε, για την αποτελεσματικότητα ενέργειας θα πρέπει βεβαίω να τα αξιολογήσουμε. Θα σας υποβάλουμε όλα τα δεδομένα στη διάθεσή σα. και συνέπεια αυτού θα είναι και ξέρω ότι πιέζει το Κοινοβούλιο ταχύτατα, χωρίς απώλεια χρόνου, πάρα χρήμα να υποβάλουμε ένα πρόγραμμα δράσης συγκεκριμένο. Δηλαδή όπως το υπολογίζω εγώ, το αργότερο αρχά του προσεχού έτου. Και για να μην ε, σα μείνει καμιά αμφιβολία ή ανησυχία. Πρέπει ο στόχο να ε, εξασφαλιστεί, να επιτευχθεί μέσα σε 10 χρόνια. Για να μην χάσουμε το στόχο του 2050 θα πρέπει να είναι δεσμευτικό ο στόχος αυτός. Και έτσι στη δική μου τη θητεία και να σας πω μια τυχαία ημερομηνία, μια πρόχειρη ημερομηνία, 2012, είμαστε διατεθειμένοι να πιέσουμε, να εργαστούμε με ταχύς ρυθμούς και στα δύο-τρία χρόνια που θα ακολουθήσουν να ετοιμάσουμε το πλαίσιο το νομοθετικό που θα είναι και δεσμευτικό, είτε προς τη μία είτε προς την άλλη πλευρά. Ο κύριος παρακαλώ. Ναι, καλό είναι το να προαναγγέλλετε εσείς ένα νέο πρόγραμμα δράσης με νομική δεσμευτικότητα, όταν όμως τα επόμενα δύο χρόνια δεν είναι καν σαφές ότι δεν μπορούμε, να, προχωρήσουμε χωρίς ένα τέτοιο πρόγραμμα δράσης. Αλλά θα προχωρήσω μια άλλη ερώτηση. Πολλά έχουν εξαγγελθεί. Με ασφάλεια βλέπουμε, ε, με βεβαιότητα βλέπουμε, ότι αντιμετωπίζουμε μαζικές αντιδράσεις ε, παγιωμένων συμφερόντων κατεστημένων συμφερόντων. Εσείς πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές τις αντιδράσεις και αντιστάσεις. Η συνεργασία σας με μη κυβερνητικέ οργανώσεις και αντίστοιχες ενώσεις πώς θα διαμορφωθεί. Απάντηση. Κύριε Βουλευτά, κύριε Μπιτικόφερ. Εμένα τα στρατεύματά μου εντό εισαγωγικών βρίσκονται εδώ σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Εσεί θα είσαστε οι σύμμαχοί μου. Εσεί θα με βοηθήσετε να διαμορφώσω την τάση η οποία θα, είναι, ε, θα έχει διαμορφωθεί σε συμφωνία όλων των πολιτικών ομάδων και θα μα πάει στο μέλλον. Και επίση σε επίπεδο Συμφουλίου και σε επίπεδο εθνική ε, ενέργειας, ε, Εθνικών Υπουργών Ενέργειας, Εθνικών Υπουργών Οικονομίας, Εθνικών Υπουργών Περιβάλλοντος θα συνεργαστώ για την διαμόρφωση αυτών των νέων προτάσεων. Και άλλωστε και η κλιματική αλλαγή και η προστασία του κλίματο και η προστασία του περιβάλλοντο δεν είναι τίποτε νέε ιδέε και προτάσει. Εδώ και 20 χρόνια περίπου είναι σαφή η κατεύθυνση προ την οποία προχωρούμε και ο, ο στόχος 20-20-20 είναι σαφώ προσδιορισμένο πιο σαφή στόχο, πιο πιστικό στόχο δεν μπορούσαμε να έχουμε. Γι' αυτό μέσα σε δύο-τρία χρόνια εγώ είμαι διατεθειμένος μέσα να, να, να διαμορφώσω δεσμευτικούς νομικά στόχους έτσι ώστε αφού η ελεύθερη αγορά και η εθελοντική δέσμευση δεν έχουν αποφέρει τους επιδιωκόμενους καρπούς ή όπου δεν τους έχουν επιφέρει, να προχωρήσουμε πιο αποτελεσματικά, πιο αποφασιστικά. Για τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις υπάρχει μια καλή συνεργασία αναπτυγμένη στις Βρυξέλλες μεταξύ των επισήμων θεσμικών οργάνων και των... Ε, ενώσεων αυτών που είναι μη κυβερνητικού χαρακτήρα και που μας συνοδεύουν στο έργο μας. Εγώ έχω προσωπική γνώση των πόσων ικανοτήτων, δεξιοτήτων και ε, προσόντων ε, μπορεί κανείς να βρει μέσα σε αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, πόσα προσόντα και ικανότητες διαθέτει το προσωπικό τους, που πρέπει να τα αξιοποιήσουμε σε μια ανοιχτή και έντιμη εταιρική σχέση. Να ακούμε τις πληροφορίες που έχουμε να μας δώσουν και να εκτιθέμεθα και στις επικρίσεις τους. Ευχαριστώ. Επόμενη ερώτηση. Κύριε υποψήφια Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την, ε, τον εφοδιασμό φυσικού αερίου από τη Ρωσία. 44% του φυσικού μας αερίου προέρχεται από αυτή την πηγή. Έχουμε το Nord Stream και 60% του φυσικού αερίου θα προέρχεται από τη Ρωσία. Και δέχεται ανοιχτά η Ρωσία ότι πρόκειται να ασκήσει πιέσεις επάνω μας και να μας χρησιμοποιήσει σαν πολιτικό μέσο αναγνωρίζετε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος αν εξαρτώμεθα όλο και περισσότερο από τη Ρωσία ως ε, προμηθευτή της ενέργειάς μας. Και αν το βλέπετε αυτό θα κάνετε κάτι για να επιταχύνετε το πρόγραμμα Αναμπούκο. Okay. Ευχαριστώ κύριε Τινιέ. Και εγώ γνωρίζω αυτές τις ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν και τις παίρνω πολύ στα σοβαρά. Γι' αυτό θα ήταν λανθασμένο να εμποδίσουμε ή να καθυστερήσουμε το πρόγραμμα Nord Stream στα πλαίσια της διαδικασίας ε, της έγκρισής του είναι η έναρξη του σχεδίου αυτού κάτι το οποίο γίνεται πια ορατό. Αλλά το να μειώσουμε την εξάρτησή μας από άλλους διάβλους μου φαίνεται ότι είναι εξίσου κατεπίγουσα και εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τον Αμπούκο και το χώρο της Μεσογείου και επίσης τη χρήση υγροποιημένου αερίου με μεταφορά με πλοία, άλλες μέθοδοι που θα μας βοηθήσουν να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τους διάβλους φυσικού αερίου. <clears throat> θα πρέπει λοιπόν για να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία μας να πράξουμε όλα αυτά ώστε να μην βρισκόμαστε σε μειονεκτική θέση λόγω της εξάρτησής μας από το ρωσικό αέριο. Ξέρω ότι οι γείτονέ μας δεν θέλουν να εξαγάγουν μονάχα φυσικό αέριο και να αποκτήσουν έτσι ε, χρήματα. Ο στόχος τους είναι με τον τρόπο αυτό να βοηθήσουν και την ανάπτυξη των χωρών τους. Αν μπορέσουμε να γίνουμε απαράγραπτοι εταίροι της Ρωσίας σε θέματα όπως η δημιουργία υποδομών, η βιομηχανία, η προστασία του περιβάλλοντος, υγειονομικά θέματα κτλ τότε αυτή η εξάρτηση θα γίνει αμφίδρομη και όχι μονόδρομος. Δεν θα έχουμε μονάχα ανταλλαγή φυσικού αερίου έναντι χρημάτων. Ε, συμπληρωματικό ερώτημα. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Στη σύμβαση της Gazprom υπάρχει ειδική ρήτρα. Η ρήτρα προορισμού όπως αποκαλείται. Καθιστά αδύνατη την πώληση φυσικού αερίου στην κοινή αγορά. Και αυτό είναι αντίθετο προς την ελεύθερη μετακίνηση, ε, διακίνηση στην ενιαία αγορά. Δεν έχουμε αμφίδρομη διαδρομή που αναφέρατε. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε έτσι την κρίση του φωτισμού σε ενέργεια. Θα κάνετε κάτι για τη ρήτρα αυτή. Κύριε Επίτροπε, έχει υπάρξει μια χρονική στιγμή που έγινε αυτή η σύμβαση που ήταν διαφορετική κατάσταση. Εγώ προσπαθώ να επιτύχω κάποια πράγματα στα οποία μπορεί να έχω περιορισμένη επιρροή, αλλά έχω κάποια επιρροή. Δεν μπορώ να επηρεάσω κάτι το οποίο έχει ήδη αποφασιστεί. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε πάντα ότι υπάρχει ο έλεγχος της συμβατότητας των συμβάσεων με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Και αν υπάρχει ε, κάποιο μειονέκτημα το οποίο προκύπτει για κράτη-μέλη τα οποία δεν συνδέονται με αυτή τη σύμβαση, είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο. Και στην περίπτωση του Nord Stream μπορούν να προκύψουν ροές φυσικού αερίου στην Ευρώπη που δεν προέρχονται από την διαδρομή του Nord Stream. Δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε εσωτερικούς διαδρόμους και διάβολους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε λογικό τίμημα για το φυσικό αέριο και ελπίζουμε ότι αυτό θα διευκολυνθεί και με την εισαγωγή, με την ε, θέση εφαρμογή του Ναμπούκο. Κύριος Μάτσιν Κίμπιτς. Ευχαριστώ. Κύριε υποψήφια επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε το πακέτο για το κλίμα και διαμορφώνουμε τώρα μια νέα πολιτική όσον αφορά την ενέργεια και την αλλαγή του κλίματος. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραματεί σημαντικότατο ρόλο σε αυτό, ανοίγει το δρόμο προς το μέλλον, αλλά πρέπει επίσης να κατευθύνει και να διαφυλάξει την εσωτερική αγορά. Πρέπει να κάνουμε την οικονομία μας πάρα πολύ ανταγωνιστική. Βλέποντας όμως τις διάφορες διατάξεις σε διάφορες νομικές πράξεις που δεχθήκαμε, βλέπω ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα για την κοινή αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Το ερώτημά μου αφορά τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσετε. Τι μεθόδους θα χρησιμοποιήσετε για να συμμορφωθείτε με τις διατάξεις του πακέτου για το κλίμα. Θα λάβετε νέα μέτρα. Ε, θα αναλάβετε νέες πρωτοβουλίες. Ούτως ώστε να μπορείτε να εγγυηθείτε την παροχή ενέργειας σε δίκαιη τιμή για όλους τους Ευρωπαίους όλα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριο Εγώ βλέπω τη δουλειά μου να αποτελεί συνέχεια του υφιστάμενου έργου του Ορεινού Επιτρόπου. Να. Ε, και πρέπει να σας πω εδώ ότι τη βρίσκω πολύ καλή και εύστοχη δουλειά, πολύ, καλή, πολύ καλά τεκμηριωμένη δουλειά αλλά ταυτόχρονα στο θέμα της ε, τεχνολογίας ενέργειας και της αγοράς της ενέργειας είναι τόσο, τόσο έντονες οι δυναμικές που ασκούνται όπως και οι δυνατότητες για αλλαγέ και μετατροπές που ασφαλώς τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να ξαναδούμε όλη την κατάσταση, θα πρέπει να κοιτάξουμε το benchmarking, του, τους προσδορισμούς δηλαδή συγκεκριμένων στόχων, και να κάνουμε ίσως ε, διαφορετικές επιλογές και ασφαλώς θα ακούσω αυτά που έχετε εσείς να πείτε, τις συμβουλές, τις υποδείξεις και τους στόχους που περιμένετε να επιτελέσω και στην εφαρμογή και στην τήρηση των υφισταμένων διατάξεων αλλά και στην διαμόρφωση νέων διατάξεων που θα είναι στο, στα καθήκοντά μου τα επόμενα χρόνια. Συμπληρωματική ερώτηση κύριε συνάδελφε. Εκπροσωπώ την Πολωνία. 95% της ενέργειάς μας προέρχεται από τον άνθρακα. Συμπληρωματική μου ερώτηση λοιπόν αφορά τους μηχανισμούς. Τι μηχανισμούς θα εφαρμόσετε σχετικά με αυτό το θέμα. Διότι η Πολωνία θα είναι μία από τις χώρες αυτές όπου τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν θα είναι τα πλέον δαπανηρά. Θα ωφεληθούμε από την αρχή της αλληλεγγύης όσον αφορά και το κόστος των επενδύσεων. Ο κύριος Έτσιγκερ. Είναι γνωστή σε μένα η ενεργειακή δομή της χώρας σας και στη δική μου την πατρίδα ο άνθρακας είτε πρόκειται για λιγνίτη είτε πρόκειται για λιθάνθρακα είτε για άλλους τύπους εισαγόμενο ή μη ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Υπάρχουν εργοστάσια λοιπόν που χρησιμοποιούν την ενέργεια του άνθρακα στην ε, Γερμανία. Η τεχνολογία Τη αποθήκευσης του οξυδίου του άνθρακα που ονομάζεται CCS θα μπορούσε να αποτελέσει την απάντηση στην ερώτησή σας. Το πώς λέει θα καταφέρουμε να ε, προχωρήσουμε τη διαδικασία της απαλλαγής από τον άνθρακα, δηλαδή της εξασφάλισης ενός κόσμου με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, πιστεύω ότι περνάει αναπόδραστα από την μέθοδο αυτή. και σε αυτό πιστεύω θα μπορούσαμε να δούμε τη δυνατότητα των επενδύσεων σε προγράμματα ερευνητικά και στην μεταφορά του διοξιδίου του άνθρακα και την ασφαλή μακροχρόνια αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Γιατί μπορεί να προσφέρει μια ε, μακροπρόθεσμη προοπτική ή ε, λειτουργία καθαρών ε, εργοστασίων που στηρίζονται στον άνθρακα για την ε, ενεργειακή τους παραγωγή σε έναν κόσμο χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Εδώ οι δομές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να μην αποβαίνουν εις βάρος των συμφερόντων συγκεκριμένων ή μεμονωμένων κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα το λόγο θα λάβει ο κύριος Αντωνέσκου. Η κυρία Αντωνέσκου, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, έχω ερώτημα που αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον πράσινο ή οικολογικό σχεδιασμό. Ποια θα είναι η πολιτική σας όσον αφορά την εφαρμογή της σχετικής οδηγίας. Τι θα προτείνετε ούτω ώστε να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της αγοράς. Υπήρξε ένα πρόβλημα με την ε, ε, διερμηνία. Μπορείτε να... Εντάξει. Μήπως μπορείτε να επαναλάβετε το, το ερώτημα. Παρακαλώ. Συγγνώμη. Micro, please. Μικρόφωνο, παρακαλώ. Deci, întrebarea se referă la eficiența energetică. Το ερώτημά μου αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον οικολογικό σχεδιασμό. Λοιπόν κύριε υποψήφια επίτροπε, ποια θα είναι η πολιτική σας όσον αφορά τον καθορισμό των εφαρμοστικών μέτρων για την εφαρμογή της οδηγίας, της οδηγίας 125 που καθορίζει το πλαίσιο για τον οικολογικό σχεδιασμό με ενδιαφέρει να μάθω τι προτίθεστε να προτείνετε για εποπτεία της αγοράς, ούτω ώστε να γίνονται σεβαστές οι προδιαγραφές. Και τι θα κάνετε ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη επικοινωνία, να ξέρουν καλύτερα επιχειρήσεις ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές. Ενημέρωση των επιχειρήσεων δηλαδή, τι σκοπεύετε να κάνετε. Κύριε πιστεύω ότι είναι πολύ καλή πολιτική πληροφόρηση της Κομισιόν. Για τα θέματα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν έχουμε έγγραφα τα οποία διατίθενται αλλά έχουμε και διασκέψεις οι οποίες ε, δίνουν δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορία σε όλους τους, ενδια... Ε, ενδιαφερόμενους. Είναι πληροφορίες οι οποίες βοηθούν στην εφαρμογή και στην αποδοχή αυτών των σχεδίων. Επομένως, η παρουσία μας σε διάφορες διασκέψεις είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους και γενικά η διεύρυνση της πληροφορίας που παρέχουμε σε όλους τους εμπλεκομένους. Τώρα, σε επίπεδο πιο λεπτομεριακό, ίσως πρέπει να μου δώσετε κάποιες εβδομάδες για να δω σε πιο λεπτομεριακό επίπεδο να ελέγξω τα θέματα της οδηγίας που έχει να κάνει με την πληροφόρηση και να δω κατά πόσο υπάρχει κάποια ανάγκη περαιτέρω βελτίωσής της. Κύριος Λάινεν. Ευχαριστώ κύριε Έτιγκερ. Νομίζω ότι έχετε αλλάξει σημαντικά, έχετε μεταστραφεί σημαντικά από την προηγούμενη αντιμετώπιση σας υπέρ της ενέργειας από το κάρβουνο και την πυρηνική ενέργεια προς τις ε, ανανεώσιμες ε, ενέργειες, αλλά είχατε ήδη σε μια προηγούμενη σας ομιλία είχατε προειδοποιήσει ότι θα ήταν επικίνδυνο να υπάρξει υπερβολική εξάρτηση από τις δημοτικές αρχές σε ό,τι αφορά την, ε, τον έλεγχο της ε, ε, πυρηνικής, ε, μάλλον της προμήθειας ενέργειας. Εσείς στο παρελθόν, στην, ε, στο κρατήδιό σας, είχατε μιλήσει ότι υπάρχει κίνδυνος υπερβολικής Ευρώπης. Τώρα μιλάτε για περισσότερη Ευρώπη, ότι είναι απαραίτητη να ξεπεράσετε τα εμπόδια τα οποία προκύπτουν από την, από την επικουρικότητα για να επιτύχετε μεγαλύτερη αποδοχή. Πώς λοιπόν μπορείτε να συμβιβάσετε αυτές τις δύο απόψεις, κύριε Έθιγκερ. όταν γίνεται ένα άλμα από ένα περιφερειακό αξίωμα, ένα τοπικό αξίωμα σε ένα ευρωπαϊκό αξίωμα και εσείς το ίδιο πράγμα έχετε κάνει. Καταρχήν, είναι απαραίτητο να έχουμε μια ευρωπαϊκή ταυτότητα στην πράξη και εξάλλου το κρατήριο από το οποίο προέρχομαι είναι διαφορετικό από άλλα κρατήδια στη Γερμανία και σε άλλες περιοχές. Εξαρτάται πάρα πολύ από την Ευρώπη γιατί βρισκόμαστε πολύ κοντά στην ε, Γαλλία. Η στρατηγική των λεγόμενων τεσσάρων κινητήρων που ξεκίνησε ο προκάτοχός μου, η στρατηγική για τον Δούναβη. Όλα αυτά μας έχουν οδηγήσει σε μια στενότερη σύνδεση με την Ευρώπη και επομένως για όλα τα θέματα που άπτονται τις ενέργειες ιδιαίτερα, εμείς ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για την σύνδεση με την Ευρώπη. Η Βάδη Βιτεβέργη δεν έχει καθόλου πυρηνικά εργοστάσια. Έχω εγκρίνει δύο νέα εργοστάσια για παραγωγή ενέργειας από άνθρακα, αλλά με πάρα πολύ σημαντικές προδιαγραφές ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά τα παλαιά εργοστάσια, τα εργοστάσια παλαιάς τεχνολογίας έχουν καταργηθεί, πάβουν να λειτουργούν και δεν υπάρχουν νέα εργοστάσια τα οποία χρησιμοποιούν το πετρέλαιο. Επομένως, όσο κανένα άλλο ε, κρατήδιο, ακολουθούμε μία οδό του μέλλοντος. Επίσης, για την βιοενέργεια και τις ανανεώσιμες ενέργειες προχωρούμε με γοργά βήματα. Η Βάδη Βιντεμπέρι σε, όχι, σε, σχέση με την ε, πυρηνική ενέργεια δεν έχει προχωρήσει προς την κατεύθυνση αυτή αλλά θέλει να υποστηρίξει τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες, γιατί από τις ενέργειες αυτές, από την ε, χρηματοδότηση των νέων ε, ενεργειών, μπορούμε να αποκομίσουμε πολλά και πρέπει να δώσουμε και την απαραίτητη υποστήριξη και στην έρευνα για τον τομέα αυτό. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια ίση σχέση με τις γαλλικές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Βάδη Βιρτεμβέργη στον τομέα της ενέργειας. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε μια εσωτερική ε, ισορροπία ώστε ένα μεγάλο μέρος των μετοχών των ενεργειακών φορέων να παραμένει στην, σε τοπικό επίπεδο στη Βάδη Βιρτεμβέργη και όχι να μεταφέρεται σε άλλες ε, χώρες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Έτιγκερ για τι απαντήσει που δώσατε μέχρι τώρα, λέει και ο Χαουτ. Θέλω πιο σαφή απαντήσεις σε δύο θέματα. Πρώτα απ' όλα, είπατε ότι ο καθορισμό παιδεγραφών θα δώσει ασφάλεια στου επενδυτέ. Εν αυτή τη ενία θα είστε πρόθυμος να πολεμήσετε μαζί μα για προδιαγραφέ, για επιδόσεις όσον αφορά ε, τις εκπομπές, όσον αφορά τι μονάδε άνθρακο, για βιοενέργεια, κριτήρια βιωσιμότητα. Ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλά πολλέ εκθέσει για τα και κατά τη βιοενέργεια. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερε εκθέσει, χρειαζόμαστε ε, κριτήρια βιωσιμότητα όσον αφορά τη βιοενέργεια. Θα είσαστε έτοιμο να πολεμήσετε για αυτά τα δεσμευτικά κριτήρια τη βιωσιμότητα. Πολύ σαφεί δύο ερωτήσει και ελπίζω να πάρω και δύο σαφεί απαντήσει. Εξάλλου, σαφεί απαντήσει έχετε δώσει μέχρι τώρα. Η βιοενέργεια δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Εξαρτάται από πού προέρχεται, πώς παράγεται και τι αλλαγή προκαλεί στο συλλογικό ε, οικολογικό ισοζύγιο. Και γι' αυτό θα πρέπει ξεκάθαρα να πούμε τι είδους βιοενέργεια θέλουμε και πώς ή ποια είναι η βιοενέργεια την οποία απορρίπτουμε και ενδεχομένως απαγορεύουμε. Και εγώ εδώ είμαι διατεθειμένος να προβώ σε επιλογές σαφείς, συγκεκριμένες και δεσμευτικές. Και βεβαίως είναι αιτιολογημένη η ερώτησή σας, αλλά δεν έχω αρχίσει ακόμη αυτή τη δουλειά. Μην ε, θεωρείτε δεδομένο ότι εγώ θα προσπαθήσω να αποφύγω τις ευθύνες που συνεπάγεται αυτό το καθήκον. Περιμένετε όταν αναλάβω καθήκοντα τι θα έχω να προσφέρω. Τώρα δεχθείτε αυτά που σας λέω ως δεσμεύσεις και επίσης για τα καθήκοντα ενός κράτους από διάφορους τομείς και ιδιαίτερα στην αυτοκινητοβιομηχανία και αρκετά νωρίς για τα οξύδια του αζότου, για τα σύγχρονα ε, συστήματα ε, καυσαερίων είδα ότι η αυτοκινητοβιομηχανία τοποθετεί τοποθετείται πολλές φορές κατά διαφοροποιημένο τρόπο όταν κάθεται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων σαν να είναι σε ένα παιχνίδι πόκερ. Έτσι λοιπόν δεν ε, πρέπει όταν ξεκινούμε αυτό το παιχνίδι του πόκερ, δηλαδή αυτές τις διαπραγματεύσεις, να κοιτάμε τι προσφέρει αυτοκίνητο βιομηχανία ή η βιομηχανία γενικότερα, αλλά να κοιτάμε πού θέλουμε εμείς να πάμε και εκεί να την υποχρεώσουμε να ακολουθήσει και να παρακολουθήσει τις προδιαγραφές που θα έχουμε ορίσει. Τη σειρά, βεβαίως και θέλω να δώσω κίνητρα και να ενθαρρύνω, αλλά τη σειρά θα την, ακολουθεί, θα την προσδιορίσουμε εμείς, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο. Φον Μπρέμπτ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, πρέπει να πω ότι είμαι κάπως απογοητευμένη. Είχατε το χρόνο να προετοιμαστείτε για αυτή την ακρόαση και θα θέλαμε να έχουμε στόχους, σαφείς στόχους και δεν μπορούμε να σας κάνουμε να μας τους παρουσιάσετε και νομίζω ότι χρησιμοποιείτε πολύ τον όρο επικουρικότητα. Το ενεργειακό μείγμα καθορίζεται βέβαια από τα κράτη-μέλη, αλλά ξέρω πάρα πολύ καλά ποια είναι τα ποσά που δίδονται σε συγκεκριμένες μορφές ενέργειας. Θέλω μία απάντηση σαφή σε σαφή ερώτηση. Είσαστε έτοιμος να προσαρμόσετε τις επιδοτήσεις ούτω ώστε να στηριχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και λιγότερο να στηριχθεί η πυρηνική ενέργεια και λιγότερο βιώσιμες πηγές ενέργειας. Ούτως ώστε να στηριχθεί η ανανεώσιμη ενέργεια και να δημιουργηθεί βιωσιμότητα στον ενεργειακό τομέα. Το κράτος θα προσδιορίσει τους στόχους ή την ε, επιλογή μεταξύ ανανεώσιμων ε, πηγών, συμβατικών πηγών κτλ. Οι διαφορές μεταξύ των κρατών δείχνουν ότι δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες. Και βεβαίως θα πρέπει και εγώ από την πλευρά μου να ε, ζητήσω να υποβληθούν εγκαίρως ε, και κατά τρόπο ε, επακριβή τα δεδομένα, τα στοιχεία για να τα μελετήσουμε. Η δουλειά, η καινούρια και κοινή δουλειά μας, θα πρέπει να σημειώσω όμως, θα γίνει αποδεκτή από τον πολίτη μόνο όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση επεμβαίνει εκεί και μόνο εκεί, με την ένταση και μόνο με την ένταση που μπορεί να προσφέρει καλύτερο αποτέλεσμα από ότι οι εθνικές αρχές. Είμαι πεπισμένος υποστηρικτής της επικουρικότητας. Και πρέπει η Ευρώπη να είναι μία διάσταση η οποία της επιτρέπει ε, να παρεμβαίνει μάλλον στη διάσταση η οποία της επιτρέπει να παρέμβει πέραν δηλαδή της εθνικής ή της τοπικής κυριαρχίας. Αυτό άλλωστε ορίζει και η συνθήκη. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε και είναι και η ευφύ επιλογή, η επικουρικότητα. Και μιλείς μόνο σε ένα, δύο, τρία χρόνια θα έχουμε μια κοινή, ένα κοινό αγώνα στο Λουξεμβούργο για κανονισμούς και οδηγίες που θα έχουμε εμείς προτείνει και εσείς εγκρίνει και όπου θα υπάρχουν πρόσφυγες ότι τάχα υπερεύει μεν τις, προ... τις ε, προδιαγραμμένες μας εξουσίες και αρμοδιότητες και ότι έχουμε προσβάλει την αρχή της επικουρικότητας. Θα έρθουν αυτές οι προσφύγες κάποια, μέρα. Και εγώ είμαι δεθμένος σε αυτόν τον αγώνα να αποδηθώ χωρίς κανένα περιορισμό, χωρίς καμία επιφύλαξη. Αλλά βέβαια, όταν ξέρω ότι όντως δεν έχω κίνδυνο να χάσω τη δίκη αυτή. Γι' αυτό και δεν θέλω να εκτεθώ σε κάποια παράβαση της αρχής της επικουρικότητας, παραβίαση της αρχής της επικουρικότητας. Παρακαλώ, συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Πότερτσνικ είπε χτες ότι πρέπει να σεβασ... γίνει σεβαστή αρχή της επικουρικότητας. Όμως αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Λαμβάνω υπόψη τη δέσμευσή σας που θέλετε να τονίσετε δηλαδή τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σημειώνω τη δέσμευσή σας αυτή. Δεν ξέρω πόσες φορές Μιλήσαμε για τη Βάδη Βιρτεμβέργη σήμερα. Δεν μιλήσαμε όμως καθόλου για τη φτώχεια, την ενεργειακή. Θα κοστίζει όλο και περισσότερο η ενέργεια και υπάρχουν κοινωνικές, κοινωνικά στρώματα που δεν θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να πληρώσουν για την ενέργεια. Τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτό το θέμα. Καθήκον μας είναι να παρακολουθούμε τις μεγαλύτερες εξελίξεις στην ενέργεια, την βασική ασφάλεια των προμηθειών για μια οικογένεια, για ένα οικοκυριό και να προσφέρουμε αυτό που χρειάζεται ένα νοικοκυριό με ασφάλεια και με οικονομία, με τιμές καλές. Αυτό είναι το καθήκον μας. Και πρέπει να παραμείνει ε, ανεκτή οικονομικά η οικονομία. Δεν μπορεί να είναι υπερβολικά ακριβή. Δεν μπορούμε να διχάσουμε δηλαδή ως προς την ενέργεια την οικονομία, την κοινωνία μας. Επίσης είναι κομμάτι του καλαφίου της νοικοκυράς η ενέργεια. Είναι ένα εμπόρευμα, ένα αγαθό το οποίο πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει αποτελεσματικά. Πρέπει ο καθένα ανεξαρτήτως της προέλευσης του τόπου διαβίωση ή των εισοδημάτων του, να έχει επαρκή ικανοποίηση των αναγκών του σε ενέργεια, όπως ακριβώς και σε ένδυση, υπόδηση, τροφή ή στέγη. Αυτό είναι κάτι το οποίο προβλέπουν, πιστεύω, όλα τα στάματα στην Ευρώπη λέμε δεν πρέπει ποτέ να κόψει κανείς το ρεύμα σε κάποιον ή το, το φυσικό αέριο ή κάνουμε συγκρίσεις των διαφορετικών ε, υποχρεώσεων που προβλέπονται για τις πολιτικές αρχές στα διάφορα, για πολιτικές αρχές στα κρατη κράτη-μέλη. Για μένα βεβαίως ίσως η καλύτερη λύση να είναι η ελεύθερη αγορά, αλλά βλέπω ότι είναι απαραίτητο οι ενεργειακές, οι επιχειρήσεις που προσφέρουν ενέργεια να υποχρεωθούν να ε, εξασφαλίσουν αυτήν την ασφάλεια, να προσφέρουν αυτήν την ασφάλεια σε προμήθεια. Συμπληρωματική ερώτηση. Αντίθετα από την προλαλήση, εγώ δεν είμαι αποκοητευμένος, αλλά πολύ ικανοποιημένο. λέει ο κύριος Λάγκεν, ε, από τα όσα μας είπατε εδώ. Ο Κλωτ Τούρμες ύστερα από πέντε χρόνια που παρακολουθεί αυτέ τι υποθέσει, πήγε δίπλα στον ε, ε, νέο κλεγέντα Βέλγο συνάδελφο για να του ψιθυρίσει αυτή τις ερωτήσει που θα σας φέρουν σε δύσκολη θέση υποτίθεται. Ε, ναι, είπε ο κύριο Λάινεν ότι αλλάξατε κασκέτο και σακάκι και ω εκ τούτου και άποψη για ορισμένα πράγματα. Μα και ο ίδιο το ίδιο έγινε. Από, λόμπι, από εκπρόσωπο των λόμπι έγινε ευρωβουλευτή. Όταν λοιπόν έχουμε κάποιον μπροστά μα, ο οποίο είναι κυβερνήτη, αρχηγό κυβερνήσεω δηλαδή τοπική ενό κρατηδίου τη Γερμανία και έχει ε, τόσα προβλήματα ήδη επιλύσει στο δικό του κρατήδιο, ξέρει να αντιμετωπίζει τι συγκρούσει, τι κρίσει και τι εντάσει. Και ρωτώ για μένα πόσο προετοιμασμένο είστε να αντιμετωπίσετε τι συγκρούσει και τι αντιπαραθέσει. Μέχρι τώρα είχαμε συζητήσεις μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Billbox και πολλούς άλλους. Εσείς πώς είστε να αντιμετωπίσετε αυτές τις συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις. Απάντηση. Εγώ βίωσα τις τελευταίες εβδομάδες μια ατμόσφαιρα ε, συλλογικού πνεύματος, ένα συλλογικό πνεύμα, ε, συνεργατικό πνεύμα μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν βλέπω λοιπόν ε, αντιπαράθεση με τους αδέλφους για την, τους αρμόδιους για την έρευνα, τις περιβαλλοντικές, ε, ε, το περιβάλλον, τη βιομηχανία, την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά εταιρική σχέση, συνεργατική σχέση. Και επίσης βλέπω ότι και εσείς στις Βρυξέλλες έχετε καταπληκτικό προσωπικό στη διάθεσή σας. Πολύ καλούς υπαλλήλους και εδώ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Γενική Διεύθυνση είναι το προσωπικό αυτό το οποίο όχι μόνο δεν επιτρέπει να ε, ταλαντευθεί η βάρκα και να μπει σε επικίνδυνα νερά, αλλά προλαβαίνει πολύ πιο νωρίτερα να συλλέξει και να διαθέσει στον ενδιαφερόμενο ε, το, το, στα στοιχεία που χρειάζεται να μελετήσει για να προετοιμαστεί, για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Εγώ δεν έχω ανάγκη από μέσα μαζική ενημέρωση για να εκφράσω τι θέσει μου, την άποψή μου σε ένα θέμα. Έρχομαι εδώ και μιλάω απευθεία μαζί σα. Αυτέ είναι οι πεπιθήσει μου. Είναι η ενέργεια, η οικονομία, η οικολογία, η προστασία ε, του πορτοφολιού του καταναλωτή, μία και ενιαία προσπάθεια. Αυτό είναι τα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνω εγώ να επιτελέσω. Ο κύριο Λάγκια για μια συμπληρωματική ερώτηση. Πολλά υπόθηκαν για τη Βάδη Βιτεμβέργη. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω και εγώ τι είδου θετικέ πτυχές θα μπορούσατε να προσφέρετε ω Πρωθυπουργό ενό μεγάλου ομοσπονδιακού κρατηδίου εφόσον επιλεγείτε. Ε, μιλήσατε για την δυσκολία στην εφαρμογή των κοινοτικών προδιαγραφών σε εθνικό επίπεδο. Από την εμπειρία σας στη διοίκηση ενός ομοσπονδιακού κράτους και τη διακυβέρνηση, τι είδους στόχους θα μπορούσατε να προσδιορίσετε για, αυτή την, ε, για την επιτεύξη αυτού του στόχου της καλύτερης εφαρμογής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Κύριε Οτιγκέρ. Εγώ θέλω να κάνω μια μικρή συνεισφορά ώστε να υπάρξει η εφαρμογή στην πράξη. Οποιοδήποτε σώμα είτε είναι τοπικό συμβούλιο, είτε είναι σε πιο υψηλό επίπεδο θεσμός, θα πρέπει να αντιμετωπίσει στόχους όπως ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης ή η αποφυγή περιττών δαπανών. Εγώ νομίζω ότι σήμερα το σύστημα των οδηγιών, οι οποίε θα πρέπει να εφαρμοστούν σε επίπεδο εθνικού δικαίου, δημιουργούν πολλές φορές προβλήματα, δημιουργούν δυσαρέσκειε. Αλλά είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε και την ε, ισορροπία των νομοθετικών αρμοδιοτήτων, διότι θεωρητικά τα λύνουν όλα τα προβλήματα οι οδηγίες, αλλά στην πράξη πρέπει να εφαρμοστούν κιόλας. Όλα αυτά οδηγούν πολλές φορές σε προβλήματα, σε επιφυλάξεις. Εγώ θέλω να σας ε, τονίσω ότι είναι απαραίτητο εν καιρό να λυθεί αυτό το πρόβλημα της έμεσης λήψης αποφάσεων σε νομοθετικό επίπεδο και να υπάρξει μια καλύτερη οργάνωση της νομοθεσίας για τα ζητήματα αυτά. Ο κύριος Λάμστορφ, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Κατά την άποψή μου έχετε σταθεί ιδιαίτερα σόφρον και πιστικός σε αυτά τα οποία είπατε και θα ήθελα να σας θέσω τώρα το πρώτο ερώτημα. Μία από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σε μια στιγμή μεγάλης κρίσης στον τομέα του, του πετρελαίου είναι και του φυσικού αερίου είναι και η συμπεριφορά ορισμένων α, φορέων. Εσείς έχετε ζητήσει να υπάρξει μια ιδιαίτερα αυστηρότερη διαδικασία για τους φορείς αυτούς. Πώς θα κινηθείτε για να εφαρμόσετε αυτές τις διαδικασίες. Να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Εάν είναι απαραίτητο να υπάρξει μια ευρωπαϊκή διαδικασία ενιαίων προτύπων για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Έτιγκερ. Είναι αριστερά σας ο κύριος Ράνστοφ. Η χρηματοδότηση και η συμμετοχή των τραπεζών σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την φερεγγιότητα δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. Αυτό δεν αφορά μονάχα τον τομέα του πετρελαίου, όπου η κρίση στον τραπεζικό τομέα είχε σαν αποτέλεσμα να τροχοπεδίσει την ε, οικονομική ανάπτυξη. Το θέμα της ε, χρηματοδότησης με επενδύσεις έχει τεθεί σε πραγματική δυσκολία, σε πραγματικό κίνδυνο. Αυτό αφορά πολλούς τομείς, όχι μόνο το τομέα του πετρελαίου και της ενέργειας. Το θέμα είναι αν οι τράπεζες θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να παίζουν το ρόλο που τους αρμόζει. Αν μπορούμε να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα υπάρξει η επαρκής χρηματοδότηση από τις τράπεζες, για να διατηρηθεί η οικονομική ανάπτυξη και να μπορούν πάντα να δίδονται οι απαραίτητες χρηματοδοτήσεις για επενδύσεις. Εγώ νομίζω ότι εδώ είναι απαραίτητο να εξασφαλίσουμε την ε, διατήρηση της ε, ικανότητας των τραπεζών. Κύριε Ράνστορφ, σας ευχαριστώ για αυτή την απάντηση. Θέλω να θέσω ένα συμπληρωματικό ερώτημα για τον νότιο διάβλο το South Stream, πώς θα ληφθεί υπόψη στην ενεργειακή δομή τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το South Stream. Για τον τομέα του φυσικού αερίου λέτε, λέει ο κύριος Σέτεγκερ. Η οδός αυτή που θα φέρει φυσικό αέριο από την Ελλάδα προς την Ιταλία. όπου φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα ε, φτηνός αυτός ο οδηγός σε σχέση με το Ναμπούκο, το οποίο είναι το αγαπημένο παιδί ίσως της ευρωπαϊκής πολιτικής, αλλά νομίζω το ο νότιος διάβλος είναι πιο προσοδοφόρος. ο διάβλος αυτός, είτε και ο βόρειος διάβλος, θα πρέπει να λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση επί τη βάση μιας εταιρικής σχέσης και ισότητος, σε ό,τι αφορά τη μεταχείριση και το κόστος. Εγώ θα προσπαθήσω στην περίπτωση του Ναμπούκο να αποφύγω τα σφάλματα τα οποία έχουν διαπραχθεί στην περίπτωση του Nord Stream. Και όλοι πιστεύω ότι έχουν συμφέρον να επιτευχθεί από αυτό. Όλοι αυτοί από οι χώρες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός, ακόμα και αυτές από δεν περνάει αλλά στις οποίες μπορεί να καταλήξει έχουν ενδιαφέρον σε κάτι τέτοιο. Μιλάμε εδώ για την Αυστρία, την ε, Ελλάδα και την Ιταλία. Είναι ένας σημαντικός χώρος, ο χώρος αυτός και εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε την λειτουργία του αγού στην περιοχή των Βαλκανίων. Βαλεάν. Κύριε Έτεγκερ, εδώ είμαι, εδώ είμαι. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα Ναμπούκο πρέπει να ξανασχεδιαστεί όσον αφορά τις διαδρομές ε, πηγές και πώς. Η κατασκευή αγωγών σε κάνει να εξαρτάσαι από, τους, από την καλή βούληση των άλλων. Τα ενεργειακά τερματικά σου επιτρέπουν να αντλήσει από διάφορες πηγές. Θα δημιουργηθούν τερματικά υγροποιημένου αερίου, θα αυξηθούν οι επενδύσεις στην Ευρώπη και πώς. Herr ε, Oettinger. Δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση μεταξύ αποθήκευσης φυσικού αερίου και διανομής με αγωγούς. Εμείς θα πρέπει να προωθήσουμε και την αποθήκευση στην Ευρώπη. Γιατί για τον Αμπούκο είναι σαφής η διαδρομή. Και το θέμα της ασφάλειας εφοδιασμού των υπολείπων κρατών που δεν βρίσκονται στη διαδρομή του Ναμπούκο είναι ένα σημαντικό θέμα. Γι' αυτό έχει νόημα να προωθήσουμε και τη δυνατότητα αποθήκευσης για να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια εφοδιασμού με όλους τους δυνατούς τρόπους μεταφοράς του φυσικού αερίου. Πολλές φορές έχουμε προέλευση από, του φυσικού αερίου από χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται σε απόλυτα δημοκρατική κατάσταση, είναι συνοδό της δημοκρατίας και εδώ αναφέρομαι σε χώρες όπως είναι το Αζερβαϊτζάν που έχουν κάθε συμφέρον να έχουν αξιόπιστες ε, σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρχει μια συγκεκριμένη παροχή ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα είναι εξασφαλισμένη. Είναι απαραίτητο λοιπόν να εξασφαλίσουμε μέσα στις συμφωνίες ότι θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί αυτή η ασφάλεια τροφοδοσίας. Συμπληρωματικό ερώτημα. Εξακολουθώ να πιστεύω ότι το Ναμπούκο χρειάζεται εκ νέου να σχεδιαστεί ίσω και οι διαδρομέ να αλλάξουν για να είναι βιώσιμο ο αγωγό. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ίσως μπορείτε να το σκεφτείτε και εσεί κατά τη θητεία σα. Ένα ερώτημα στο τέλο. Τι σκέφτεσαι για το τρίγωνο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ενώσης, Ουκρανίας και Ρωσίας όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική. Ένα τρίγωνο αγάπης αν θέλετε. Κύριε Όσο επικίνδυνα και τραγικά να ήταν τα πράγματα όπως εκδηλώθηκαν τα τελευταία χρόνια, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορέσει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της με έγκαιρη προειδοποίηση, με ενεργό δράση, με σκληρή μερικές φορές ε, γλώσσα προς το Κίεβο και προς τη Μόσχα και έτσι μπόρεσε να αποφύγει ε, τις χειρότερες ζημιές. Απέδειξε δηλαδή την ικανότητά της να διαχειρίζεται τέτοια προβλήματα. Αυτό που μπόρεσε να επιτύχει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μόνα του το καθένα ξεχωριστά, δεν θα μπορούσαν να το επιτύχουν. Μέγιστη απόδειξη της σημασίας και της αξίας Ευρωπαϊκής Ένωση και για τον συνάδελφο Πίμπαλξ. Έγκαιρο σύστημα Έγκαιρο προσδιορισμό προσδιορισμός ε, ε, ε, έγκαιρη, ενημέρωση καθήκον έγκαιρης ενημέρωσης, κοινοποίησης και από τον περσινό Ιανουάριο μέχρι τώρα βλέπουμε ότι μπορέσαμε να αποκλείσουμε κάθε είδους επιθέσεις, να μην τολμήσει κανείς δηλαδή να κάνει τέτοιου είδους επιθέσεις βάρος μας. Και πρέπει από την άλλη πλευρά να επαληθεύσουμε για τα κράτη ενδεχομένω, για μας όλους, εάν οι προθεσμίες που θα ορίσουμε για την ασφάλεια των ε, ενεργειακών μας προμηθειών που χρειαζόμαστε για την παραγωγή μας θα είναι 60 κονταήμερη ή 90 κονταήμερη ε, περίοδος. Για δε το μέλλον βλέπω ότι ένα κράτος θα πρέπει να είναι σε θέση όταν δεν έχει αρκετές ποσότητας ενέργειας στη διάθεσή του να ζητεί τη βοήθεια ενός άλλου κράτους και να την εξασφαλίσει. Το ίδιο και για μια επιχείρηση ενδεχομένως, δηλαδή όλοι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δρούμε αλληλέγγυα, να προσφέρουμε χείρα βοηθείας την ώρα που τα πράγματα πάνε στραβά για κάποιον η διαδικασία που προέκυψε τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι είχε τραγικέ διαστάσει, δραματική μάλλον ε, διάσταση και διαμόρφωση, αλλά μπορέσαν όλοι να σταθούν όλοι στου άλλου αλληλέγγυοι. Ο επόμενος ομιλητή, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Έτιγκερ. Ευχαριστώ για τι πιστικές πληροφορίε και τι ιδέε που παρουσιάσατε μέχρι τώρα. Συμφωνώ με τα περισσότερα από αυτά που είπατε, εκτός ίσως την πολιτική σα για την πυρηνική ενέργεια αυτό βέβαια είναι πάντα αμφισβητούμενο θέμα. Για μια στιγμή πάμε στο μέλλον. Θα εκτιμούσα την άποψή σας και τα οράματά σας όσον αφορά τις μελλοντικές εξελίξεις ε, ε, εναλλακτικών πηγών ενέργειας βάσει νέων προχωρημένων τεχνολογιών. Τα κινητήρε κινητήρες υδρογόνου που θα χρησιμοποιηθούν κυρίως τα αυτοκίνητα. και κάτι που θα είναι πιο σημαντικό στο μέλλον, οι αντιδραστήρες σύνδεξης. Αντί από την καύση ορυκτών καυσίμων, οι διαδικασίες αυτές δεν παράγουν διοξίδιο του άνθρακος ούτε αέρια του θερμοκηπίου. Επίτροπε, υποψήφια επίτροπε, θα εντάξατε την προώθηση αυτών των νέων τεχνολογιών στο πρόγραμμά σας, τουλάχιστον όσον αφορά την έρευνα και την καινοτομία. Ή προς το τέλος της θητείας σας Δεν ακούγεται ο μιλητή λόγω σημάτων του που πατάει το καμπανάκι ο πρόεδρο. Λυπούμαστε. Υπάρχουν πολλοί τομεί <clears throat> στου οποίου είναι αρκετά μεγάλε οι επιχειρήσει για να προχωρήσουν σε έρευνα. Σε άλλες περιπτώσεις το ρόλο αυτό πρέπει να το κάνουν τα εθνικά ερευνητικά ιδρύματα. Είναι περιπτώσεις όμως τομέων του επιστητού που είναι τόσο, πλή, που μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Και ο τομέας ενέργειας είναι ένας χώρος στον οποίο όλοι οι ευρωπαϊκοί εταίροι θα πρέπει να συμμετάσχουν στην έρευνα. Για μένα λοιπόν το θέμα της ερευνητικής εργασίας στην ενέργεια είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να δώσουμε σημαντικά περισσότερα μέσα στην έρευνα μετά από την πετρελαϊκή κρίση στη δεκαετία του 70. Τα ευρωπαϊκά κράτη έδωσαν πολύ μεγαλύτερα κονδύλια για την ενεργειακή έρευνα από ό,τι στο παρελθόν. Περισσότερα λοιπόν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν την μελλοντική παραγωγή ε, σε συνθήκες αποδοτικές. Υπήρξαν πολλά προβλήματα, προγράμματα λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και υπάρχει και μια καλύτερη διαδικτύωση των εργαζομένων στην έρευνα για την ενέργεια. Υπάρχουν ε, ιδρύματα όπως το Φρανχόφερ, το Max Planck στη χώρα μου που παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτά και έχουμε δημιουργήσει και ένα κέντρο ποινικής έρευνας στην Καλσρούη ε, που αποτελεί ένα έδος φάρου για την έρευνα στην πυρηνική ενέργεια και το οποίο συνδέεται πια πάρα πολύ στενά με τα πανεπιστήμια μας. Έχουμε λοιπόν μια δομή η οποία μοιάζει πια με το MIT στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει αυτό να κάνουμε για να έχουμε τις δομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι οποίες θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη έρευνα στον τομέα της ενέργειας. Θέλουμε λοιπόν να μην μας ξεπεράσει κανένα άλλο τμήμα του κόσμου σε ταχύτητα και σε ικανότητα να αναπτύσσουμε νέες ενεργειακές τεχνικές. Αυτό είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα της δικής μου εργασίας και των αρμοδίων για την έρευνα στην ε, Νέα Κομισιόν. Παρακαλώ για συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ίσως θα πρέπει να το συζητήσουμε εκτενέστερα στο μέλλον το θέμα να επιστρέψουμε στην εξάρτηση χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε ενεργειακές πηγές από τη Ρωσία, κυρίως στον φατοφυσικό αέριο. Σε κάποιε περιπτώσει θα είναι το 100% η εξάρτηση, όπω στη χώρα μου, στη Σλοβακία. Στην περίπτωση χωρών κεντρική Ανατολική Ευρώπη είναι ανησυχητικό το φαινόμενο. Αν δούμε την, την άσχημη εμπειρία τη περσινού Ιανουαρίου στον αυτοφυσικό αέριο βλέπουμε ότι υπάρχουν πτυχέ οικονομικέ και πολιτικέ. Ποια πτυχή από αυτέ θεωρείται σαν την σημαντικότερη σαν την κινητήρια δύναμη για να βοηθήσει να βρούμε μια λύση για να μειωθεί η ρωσική επιρροή σε ενεργειακά θέματα. Νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε καλό συμβιβασμό τελικά μεταξύ πολιτικής και οικονομίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σέτσιγκερ παρακαλώ για να απαντήσω. Θα αναλάβω, και αυτό δεν είναι γνωστό για την κοινή γνώμη, ότι θα, το θέμα βλέποντας ποια είναι τα κράτη από τα οποία, τα οποία έχουν μηδενική εξάρτηση από τη Ρωσία, Ρωσία και τα άλλα τα οποία μερικέ φορέ έχουν μέχρι και 100% εξάρτηση. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τη διαδικασία τη εκδήλωση ελληνική και με την εσωτερική αγορά. Δεν θα μείνει κανεί μόνο του εκτεθειμένο σε πιέσει ή σε στέρηση. Αυτό είναι το δεδομένο το οποίο εγώ μπορώ να αξιοποιήσω. Έχοντας βέβαια γνώση του γεγονός ότι είναι ιστορική εξέλιξη, έχει ιστορικούς, ιστορικές ρίζες αυτή η εξέλιξη, αλλά ταυτόχρονα για την Ευρώπη εμείς διεκδικούμε την, την ελευθερία και την ανεξαρτησία στη δράση μας ως πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα της πολιτικής μας διαμόρφωσης. Και μια τελευταία λέξη αυτό, εγώ την ε, Ρωσία με κάθε ανεξαρτησία βέβαια απέναντί της τη βλέπω ως ένα πολύ σημαντικό εταίρο. Αλλά αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και την υποχρέωση για την ανάπτυξη στενών δεσμών ε, με όλα τα κράτη έτσι ώστε η Ρωσία ποτέ να μην είναι σε θέση να αξιοποιήσει εις βάρος των κρατών αυτών ε, την θέση της. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λέει κύριο Κύριε υποψήφια επίτροπε, ευτυχώς ή δυστυχώς απαντήσατε όλες τις ερωτήσεις που είχα ετοιμάσει. Και γι' αυτό θα αναφερθώ στην αλληλεγγύη. Διότι η αλληλεγγύη μεταξύ των 27 κρατών μελών είναι ζωτική σημασίας για να εξασφαλιστεί ο ασφαλής εφοδιασμός, ο ενεργειακός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχοντας αυτό υπόψη, σε περίπτωση κρίσεως όσον αφορά την παροχή φυσικού αερίου, πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί μια λύση, να δημιουργηθούν αποθήκες ενέργειας σε διάφορες περιφέρειες, περιοχές για να δημιουργηθούν στατηγικά αποθέματα χρησιμοποιώντας το πρότυπο, πρότυπο δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως κάνουν με το πετρέλαιο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μία απάντηση για την αντιμετώπιση της εξάρτησης είναι η αποθηκεύση. Και αυτό ισχύει για όλους τους ενεργειακούς πόρους. Είναι μια απάντηση σε όλους στα προβλήματα εξάρτησης από όλους. Αν θέλουμε παραδείγματος χάρη να εξασφαλίσουμε την παραγωγή από ε, ανανεώσιμες ενέργειες, έχουμε παραδείγματος την ε, υδροηλεκτρική ενέργεια και τη χρήση της για τις μεταφορές ή στις Άλπεις υδροηλεκτρική ενέργεια και επίσης τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας από από αιωλική ενέργεια, να μπορούμε να μετατρέψουμε σε μορφές που μπορούν να αποθηκευθούν, όπως είναι παγκοσχάρι, σε δεξαμενές ύδατος. Ε, Όλα αυτά ισχύουν λοιπόν και για το φυσικό αέριο, αλλά και την δυνατότητα των ενεργειών που είναι ανανεώσιμες να αποθηκεύονται με μια μορφή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στη συνέχεια. Ε, συμπληρωματικό ερώτημα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συμπληρωματική ερώτηση. Η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτηρίων είναι το θέμα της ερώτησης. Διότι δεν έχουμε συγκεκριμένα κονδύλια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως για αυτού του είδους τη δραστηριότητα. Λοιπόν κύριε υποψήφιε επίτροπε θα ήταν δυνατόν κατά τη διάρκεια του επομένου προπολογισμού και των σχετικών διαπραγματεύσεων από τα διευθυντικά ταμεία και τα επιχειρησιακά προγράμματα να υποστηρίξετε κάποιοι πόροι να μεταφερθούν για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων. In ähm, Σε θέματα προπολογισμού εσείς αποφασίζετε. Άρα θα εξαρτηθούν τα πάντα από το τι λεφτά θα μπορέσουμε να αποσπάσουμε από τα εθνικά κράτη, από το ΑΕΠ τους, γιατί ίσως να μην υπάρχει πρόθεση, καλή διάθεση για μεγάλα άλματα. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι το θέμα της ενέργειας σημαίνει θα πρέπει να ασκήσουμε στο βαθμό που μπορούμε την πυθό μας έναντι των εκπροσώπων της εθνικής πολιτικής. Και ταυτόχρονα θα πρέπει και να μετατοπίσουμε τις προτεραιότητες ενδεχομένως. Θα έρθει η στιγμή να εξετάσουμε και αυτό το θέμα και στη συζήτηση, στη λειτουργία, στις επιλογές θα έρθει η στιγμή να δώσουμε περισσότερα κονδύλια στον προπολογισμό, ειδικά για την ενέργεια. Πιστεύω δε ότι η αξιοποίηση υφισταμένων προγραμμάτων, διαρθρωτικών υφισταμένων προγραμμάτων, περιφερειακών υφισταμένων προγραμμάτων, θα μπορούσαμε να προβλέψουμε κίνητρα, όθηση που να στοχεύει ειδικότερα στην ενέργεια και με τον συνάδελφο Χάν θα πρέπει να συζητήσω εάν η ενεργειακή πολιτική μπορεί να βρει τη θέση της ε, και περισσότερους πόρους για τους στόχους μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, συμφωνώ με εκείνους τους συναδέλφους που είναι ικανοποιημένοι από την όλη προετοιμασία που κάνατε για τη συνεδρίαση. Πολλές από τις απαντήσεις σας ήταν σωστές, πολύ έξυπνες και είναι πολύ σημαντικό διότι οι απαντήσεις ήταν ειλικρινείς. Απαντήσατε σε πολλά σημεία που με ανησυχούσαν σχετικά με τον εφοδιασμό, τη διασύνδεση μεταξύ των περιοχών κλπ αλλά θα ήθελα να περάσω σε ένα συμπληρωματικό ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξέρω πώς θα λύσετε το εξής πρόβλημα. Το πρόγραμμα σύνδεσης Λιθουανίας και Πολωνίας με φυσικό αέριο δεν βρίσκει επενδύσεις διότι ε, δεν υπάρχουν επαρκή σπόροι, αλλά είναι κάτι απαραίτητο να γίνει για θέμα ασφαλείας εφοδιασμού. Θα βρείτε για τέτοιου είδους διασυνδέσεις και τέτοια προγράμματα χρηματοδότηση. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Εμείς θέλουμε να δώσουμε πάντα τον κύριο το θέμα αυτό πρέπει να δοθεί κυρίως από τον Επίτροπο Οικονομίας. Αλλά και για μένα επίσης είναι σημαντικό να δώσουμε μια απάντηση στα ερώτημα αυτά. Όταν είναι περιορισμένες οι δυνατότητες των ε, κρατών αυτών και δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια οδό διέλευσης του φυσικού αερίου ή οποιοδήποτε άλλου ενεργειακού πόρου, θα πρέπει τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίσει την χρηματοδότηση, παραδείγματος χάρη, μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η οποία θα πρεπει τοτε η ευρωπαικη ενωση να εξασφαλισει την χρηματοδοτηση παραδειγματο μεσω τη ευρωπαικης τραπεζα επενδυσεων η οποια θα κανει τι απαραίτητε ενέργειες για να δώσει εγγυήσει σε <clears throat> ευνοϊκά επιτόκια για τις επενδύσεις αυτές. Αλλά αυτό μόνο σε τελική ανάλυση. Ο στόχος μας θα πρέπει να είναι η περιοχή της Βαλτικής να ενσωματωθεί στον ευρωπαϊκό χώρο ενέργειας και να μπορέσει αυτό να γίνει μέσα στο, στην επόμενη δεκαετία. Συμπληρωματικό ερώτημα. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω απλώς για την απάντησή σας. Ευχαριστώ κυρία Χέρτσοκ. Και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω κοντά μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι και εγώ που είμαι ξανά εδώ σε αυτή την Επιτροπή και διαβεβαιώνω τον υποψήφιο Επίτροπο ότι ποτέ δεν θα μείνω χωρί ερωτήσει όσον αφορά το ενεργειακό. Κύριε Επίτροπε, υποψήφιο Επίτροπε, θα είστε υπεύθυνο για ενεργειακή έρευνα στο μέλλον και πρέπει να βασιστείτε στη, στο σχέδιο στρατηγικής, στρατηγικό σχέδιο τεχνολογίας και θέλουμε να ηγηθείτε στον τομέα αυτό. Πρέπει να εστιαστεί εκ νέου η έρευνα ε, για την ενέργεια σε έρευνα που μπορεί να απευθύνει και στη βιομηχανία που δημιουργεί θέσει απασχόληση. Και μα βοηθά να πετύχουμε του στρατηγικού στόχου. Όσον αφορά λοιπόν το σχέδιο αυτό στρατηγικό για την ενέργεια, δημοσίευσε τον Οκτώβριο 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ανακοίνωση που περιγράφει τι οικονομικέ απαιτήσει. 50 δισεκατομμύρια ευρώ κατά την επόμενη δεκαετία για την ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών με χαμηλέ εκπομπέ άνθρακα για το μέλλον. Το ερώτημά μου είναι απλό. Τι θα κάνετε για να μαζέψετε τα 50 δις Πώς θα τα καταφέρετε λοιπόν να μαζέψετε αυτά τα χρήματα, αυτό είναι το ερώτημα. Κυρία Βουλευτή, η δουλειά μου θα είναι να συζητήσω με την αρμόδια για την έρευνα συνάδελφο, πάντα σε σεβασμό των ε, διαφορετικών μας ε, αρμοδιοτήτων, των αρμοδιοτήτων μας και με τον υπεύθυνο για τα θέματα του προϋπολογισμού, να συζητήσω τα θέματα αυτά, να, να προχωρήσω στην μελέτη της υπόθεσης. Αυτό θα είναι το πρώτο καθήκον. Και μετά, στα προσεχή χρόνια, καθήκον μου είναι, κατά με, το να προετοιμάσω για τις μελλοντικές αποφάσεις σχετικέ με τον προϋπολογισμό, τις πλειοψηφίες, την υποστήριξη που χρειάζομαι. Επίσης, τα ερευνητικά προγράμματα θα προσπαθήσω να τα συνδυάσω στο μέγιστο δυνατό βαθμό με τα εθνικά και περιφερειακά ερευνητικά προγράμματα όπως αυτά αναπτύσσονται και μάλιστα υπάρχουν σε μεγάλες, ε, υπάρχουν πολλοί άριθμα στα κράτη-μέλη και στις περιφέρειες. Επίσης, θα κοιτάξω την ενεργειακή οικονομία, την οικονομία της ενέργειας, την τεχνολογία της ενέργειας, την οικονομία εκείνη η οποία παράγει νέα τεχνολογία για την ενέργεια. Δηλαδή, θέλω να δεσμεύσω και τις μεγάλες ερευνητικές ε, μονάδες, τα μεγάλα ερευνητικά κέντρα, που θα μου δίνουν αποτελέσματα της έρευνάς τους και τα οποία εγώ θα μπορώ να διαβιβάσω στη συνέχεια, να διοικητεύσω στην οικονομία, με συγχρηματοδότηση ενδεχομένω, χάρη στι καλέ πρακτικέ του εφαρμογέ, για να αποφέρουν εις όφελος των πάντων. Με εταιρικέ σχέσεις των ερευνητών που δρούν στο δημόσιο χώρο ή σε συγκεκριμένες εταιρικέ σχέσεις. Και εδώ νομίζω ότι μπορούμε να συγκεράσουμε, να συνενώσουμε τις δυνάμεις των μεν και των δε και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Συμπληρωματική ερώτηση, κυρία Χέρτσοκ. Σας ευχαριστώ, κύριε Έτιγκερ. Πρέπει να θυμόσαστε ότι αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σας, θα σας υποστηρίξει. Η Επιτροπή μας σας υποστηρίξει στον αυτά τα μέτρα. Θα πρέπει να ετοιμαστεί το σχέδιο δράσεως ε, μέχρι, μεταξύ 2010-2014. Τι σκοπεύετε να κάνετε, τι προστιθέμενη αξία ε, θα, θα προστιθέμενη αξία θα δώσετε στο κείμενο που βγήκε από την Ερηνή Συνοδοκορυφής. απάντηση. Θα... Εφόσον βεβαίως ε, μας ε, επικυρώσετε και μας καλέσετε να αναλάβουμε καθήματα, τα καθήκοντα, στην πρώτη συνεδρίαση θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι έχει να συμβάλει στην Ερηνή Σύνοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμένα η δική μου συμβολή θα είναι ο ρόλος του, του, της ενέργειας και της προστασίας του κλίματος, των κλιματικών αλλαγών θα είναι πάνω από όλο αυτό. Μέσα με τα υπόλοιπα θεματικά τα οποία θα προκύψουν εν πορεία. Και μετά από εκεί και πέρα τα πράγματα προχωρούν αρκετά γρήγορα. Από την ανάληψη καθηκόντων την 1η Φεβρουαρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάποιοι διαβλέπουν μειονεκτήματα. Εγώ διαβλέπω πλέον διότι μπορώ να έχω περισσότερο χρόνο για επικοινωνία και ατύπως ήδη σας προσκαλώ σε επικοινωνία, σε επαφή τον Φεβρουάριο για να ακούσω τι έχετε εσείς να ζητήσετε ως θεματολογία σε αυτήν την έρηνη σύνοδο. Πιστεύω ότι και η Ισπανική Προεδρία, η νέα αυτή Προεδρία, έχει υψηλές φιλοδοξίες προσδορίσει και για το θέμα της ενέργειας και νομίζω ότι μπορούμε την ευκαιρία το Φεβρουάριο να την αδράξουμε ώστε να μπορούμε να προσδορίσουμε τις σωστές και για σας κατευθύνσεις. Ευχαριστώ. Κύριος Πίπερ. Κύριε Έτσιγκερ, έχουμε ε, δει από πλευρά σας οράματα και ευφύς επιλογές. Αλλά αν δεν κάνω λάθος το παιχνίδι, αυτό το σκάρτ το οποίο παίζεται, ο κατάλογος των αποτελεσμάτων, το φύλλο αποτελεσμάτων έχει μόνο μαύρο και κόκκινο να συμπληρώσει κανείς, δεν έχει γκρίζο ή ενδιάμεσα χρώματα. Θα ήθελα λοιπόν συγκεκριμένους στόχους για το 2050 οι διάφοροι άσοι, τα διάφορα πλεονεκτήματα που έχουμε στη θέση μας αυτή τη στιγμή είναι οι οικολογικοί φόροι, τα συστήματα τα αυστηρά για την αποθήκευση, ε, η αποτελεσματικότητα της ενέργειας, ήδη ο πολίτης κατευθύνεται στην, στην καθημερινή του ζωή προς την πρακτική αυτή. Ερωτώ λοιπόν, θέσεις εργασίας, κοινωνικά προβλήματα, ε, οι ομάδες ευάλωτες κοινωνικά μπορούν να συμπεριληφθούν μέσα σε αυτό το μεγάλο όραμα και τη στρατηγική που μας περιγράψατε για να φτάσουμε σε αυτό το 20%. Απάντηση. Φυσικά και πρέπει να συζητήσουμε ε, με ανοιχτά χαρτιά για να βρούμε την απάντηση στην ερώτησή σας. Η στρατηγική πρέπει να προσδιορίζει αυτόν τον στόχο. Και πιστεύω ότι το να προσδιορίσουμε καθήκοντα και στόχους συγκεκριμένου για τη βιομηχανία έχει νόημα μόνο εφόσον τους στόχους μπορεί να τους εξασφαλίσει, να τους επιτύχει η βιομηχανία και ταυτόχρονα αν μπορούμε να διαφυλάξουμε και τις θέσεις εργασία στη βιομηχανία. Δηλαδή αν ορίσουμε έναν πολύ στόχο που θα έχει ένα αποτέλεσμα να ε, φύγουν όλοι από την Ευρώπη ή να χάσουμε τις θέσεις εργασία, ε, τότε η προστασία του κλίματος θα έχει αποτύχει ο στόχος. Θα έχει, ε, θα έχει επιλεγεί λάθος μέσον για το στόχο αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να μιλήσει με απόλυτους όρους για το ποια θα είναι η κατάσταση το 2020 το 2030 σε ολόκληρο τον κόσμο, αλλά και σε ποιο βαθμό θα μπορέσει να προχωρήσει η αποδοχή, ο βαθμός αποδοχής καλύτερα των στόχων μας από τον πολίτη και την πολιτική στα επόμενα χρόνια. Αναλόγως λοιπόν θα πρέπει να προχωρούμε σε διορθωτικές κινήσεις. Όχι μόνο δηλαδή το step by step, βήμα το βήμα, αλλά ταυτόχρονα έχοντας πάντοτε ένα στόχο στο, στο νου μας, να διορθώνουμε την πορεία μας όσο και εφόσον χρειάζεται. Εγώ τίνω προς τα φιλόδοξα οράματα περισσότερο και είμαι διατεθειμένος να δεσμευτώ και σε φιλόδοξα οράματα. Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται και όλοι μας να συμμετάσχουμε και να παραμείνουμε δεσμευμένοι, στρατευμένοι σε αυτόν τον αγώνα για να έχουμε καλά αποτελέσματα και να έχουμε την ευελιξία να διορθώσουμε την πορεία μας όταν χρειαστεί. Για να μπορούμε να έχουμε καλά προγράμματα είτε δεκαετίας, είτε εικοσαετίας ή και τέσσερα κονταετίας ακόμα. Ένα ερώτημα συμπληρωματικό για τα επόμενα πέντε χρόνια, κύριε Έτογκερ. Η δική σας προσωπική στόχη που έχετε θέσει για τον εαυτό σας. Πού μπορούμε να βρισκόμαστε μετά από πέντε χρόνια, κατά την άποψή σας. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανακτήσει την βιομηχανική της ανταγωνιστικότητα και μέσα από αυτό υπάρχει μια ευκαιρία στην τομέα της ενέργειας να προχωρήσουμε προς μια αηφόρο ενέργεια και να έχουμε νέες τεχνολογίες οι οποίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον στον τομέα της ενέργειας. Και γι' αυτό σκέφτομαι για την πράσινη ενέργεια αφενός, αλλά και τις ευφυείς τεχνολογίες για την διαδικτύωση της ενέργειας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικοί παράγοντες και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε μια νέα αντιμετώπιση η οποία θα είναι πιο στοχευμένη στην ανταγωνιστικότητα αφενός και αφετέρου στην αηφόρο. Όλα αυτά θα είναι αποφασιστικά επομένως μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια και φυσικά θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και τις δυνατότητες που μας δίνει η συνθήκη της Λισαβόνας για να προωθήσουμε περισσότερο τους δύο αυτούς τομείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας Πάσκο. Κύριε Επίτροπε, κύριε υποψήφιοι Επίτροπε, μιλήσατε για την αναγκαία διαφοροποίηση της ενέργειας για το ενεργειακό μείγμα. Εδώ είμαι, με βλέπετε. Στο οποίο θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες επιλογές. Υπάρχει μεγάλο δυναμικό στον τομέα της ενέργειας και αυτό είναι η υδροηλεκτρική ενέργεια. Μιλήσετε για μια μεγάλη στρατηγική των τεσσάρων κινητήρων. Ερωτώ λοιπόν, έχετε κάποια συγκεκριμένη ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο τα δυναμικό που προσφέρει η υδροηλεκτρική ενέργεια. Απάντηση. Η στρατηγική του Δούναβη είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά με ε, ενδιαφέρει, ένα έργο πνοής για μένα, διότι ξεκινάει από την πατρίδα μου, ένα, από την ιδιαίτερη μου πατρίδα βέβαια, ε, και αναπτύσσεται γύρω από τα ιδρυτικά τρία-τέσσερα κράτη-μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ο Δούναβης έναν, μίαν οδό όχι μόνο υδάτινη, αλλά και πολιτιστική, αλλά και ιστορική, αλλά και οικονομική και, ε, περιβαλλοντική. Γι' αυτό βλέπω λιμένες, γι' αυτό βλέπω ε, φορτίο, μεταφορά φορτίου μέσα από το υδάτινη οδό και όχι μόνο βέβαια τον ε, Δούναβη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στο δούναβη πάνω δεν είναι μόνο οι γερμανικές πόλεις, αλλά είναι και η Βουδαπέστη και το Βελιγράδι. Το ίδιο ισχύει και για την υδροελεκτρική ενέργεια. Στρατηγικό σχέδιο για την αξιοποίηση του Δούναβη για την ε, προσαρμογή του έτσι ώστε να είναι κατάλληλος για πλεύση σε, όλες σε όλο του το μήκος, έτσι ώστε να ε, απορροφήσει μέρος του φορτίου από τους οδούς, αλλά και για την υδροελεκτρική ενέργεια νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε τις λύσεις. Απάντηση. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. Ναι. Είπατε ότι μπορέσαμε να, αξιοποιήσουμε, να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ενεργειακή κρίση και από πέρσι δεν είχαμε πρόβλημα διελκυστίνδα με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Η σλοβακική κυβέρνηση όμω βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση γιατί χρειάστηκε να ε, περάσει μια μεγάλη περίοδο χωρί φυσικό αέριο όταν ευρωπαϊκά κράτη τα οποία είναι, ε, έχουν στην κατοχή τους αποθηκευμένο φυσικό αέριο δεν ήταν διτεθειμένα να το μοιραστούν. Οι μεγάλες επιχειρήσεις καλύτερα. Έναντι αυτών των μεγάλων επιχειρήσεων λοιπόν που δεν έδειξαν αλληλεγγύη, εσείς πώς θα στέκεστε. Απάντηση. Η ενέργεια είναι βέβαια και προϊόν, αγαθό στην αγορά, αλλά και ένα αγαθό ε, κοινό, ένα αγαθό απαραίτητο για τους πάντες και ως εκ του μπορούν να ισχύουν οι κανόνες της αγοράς, της ελεύθερης αγοράς, αλλά όχι καταχρηστικά. Και γι' αυτό πρέπει να προσδιοριστεί ε, ένα σύνολο κανόνων πιο αυστηρών για τον τομέα του εμπορίου σε ενέργεια. Όταν ένα κράτος λοιπόν μπορεί, να μπορεί αποδεδειγμένα να ε, κινδυνεύει από εξάρτηση, δηλαδή από αποστέρηση από προμήθεια ή από εφοδιασμό στις απαιτούμενες ποσότητες ή μορφές ενέργειας, τότε οι κάτοχοι αποθηκευμένων ε, μορφών ενέργειας θα πρέπει να είναι η υποχρεωμένοι να τους υποδειχθεί η υποχρέωση για ε, διάθεση της αποθηκευμένης αυτής ενέργειας για το κοινό καλό. και να ε, υπάρξει αυτή η υποχρέωση για διάθεση στον λόγο κράτος των απαραίτητων όγκων. Εδώ η ασφάλεια σε ενέργεια πρέπει νομίζω να ε, εξεταστεί με ιδιαίτερη ευαισθησία. Γιατί είναι ένα αγαθό απαραίτητο όπως κάθε άλλο βασικό αγαθό στη ζωή του ανθρώπου. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε κύριε Έτιγκερ. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ότι τον 21ο αιώνα η ενέργεια είναι εξίσου σημαντικός πόρος όπως τα τρόφιμα και το νερό. Όμως όταν μιλάμε για τον ασφαλή εφοδιακό, ενεργειακό εφοδιασμό το θεωρούμε τεχνικό θέμα και δεν αναφερόμαστε στο κόστος ε, της ενέργειας. Η απελευθέρωση των αγορών δεν ήταν κάτι υποφελές για όλους, όπως για τη χώρα μου την Ουγγαρία. Οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη, ενώ οι προμηθευτές ενέργειας ε, τσέπωσαν τεράστια κέρδη. Και εδώ το ερώτημά μου. Εάν πιστεύετε στην κοινωνική δικαιοσύνη όσον αφορά τις κοινοφελείς υπηρεσίες, τότε τι πρακτικά μέτρα θέλετε να εφαρμόσετε για να μειωθεί η ενεργειακή φτώχεια. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιο επίτροπε. Όλοι μας θέλουμε να έχουμε ένα σπίτι το οποίο θερμαίνεται, σε στο νερό, βασικές ανάγκες να καλύψουμε λοιπόν και να έχουμε τις συνθήκες αυτές οι οποίες ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Χωρίς ενέργεια δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε αυτές τις βασικές ανάγκες. Επομένως, τα μέτρα μας να έχουμε οδούς μεταφοράς ενέργειας, να συμπληρώσουμε την εσωτερική αγορά, να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα, θα πρέπει να οδηγήσουν στο το τίμημα της ενέργειας να είναι προσιτό και προσβάσιμο για όλους τους καταναλωτές. Πρέπει λοιπόν η ευρωπαϊκή πολιτική να μην ξεχάσει το θέμα της προσιτότητας των τιμών ενεργείας. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο αξίζει να αντιμετωπιστεί και με μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση και θα πρέπει <clears throat> να υπάρξει και ένας κώδικας συμπεριφοράς για τις εταιρείες που περιορίζει τη δυνατότητά τους να αποστερούν τον καταναλωτή από την ε, παροχή ενέργειας. Εγώ πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει μια διασύνδεση. Στην Γερμανία υπάρχει υποχρέωση στα τραπεζικά ιδρύματα να δίνουν λογαριασμούς τραπεζικούς σε όλους και όχι να επιλέγουν σε ποιον δίδουν λογαριασμού και σε ποιον όχι. Πρέπει να υπάρχει μια αντίστοιχη υποχρέωση για τι εταιρείε ενέργεια. Να πρέπει να είναι υποχρεωμένε να δίνουν ενεργειακά προϊόντα σε όλου. Η φορολογία τώρα, η διάρθρωση των τιμών, η ρύθμιση, η ρύθμιση της αγοράς θα πρέπει λοιπόν να λάβουν υπόψη αυτό το πραγματικό καθήκον να υπάρχει προσβασιμότητα σε όλους, για όλους σας στην ενέργεια και να εξασφαλίσουν αυτό το στόχο. Συμπληρωματικό ερώτημα. Έχω στα χέρια μου το πιο πρόσφατη έκδοση του Finance Plat που το έλαβα χτες και βλέπετε στην πρώτη σελίδα τα συμπεράσματα ενός τραπεζίτη. Η κοινωνική οικονομία είναι σαν βασική έννοια δεν έχει αποτύχει. Αυτό είναι ο τίτλος. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δράσετε συγχρονιζόμενος με την κοινωνία και τις επικρατούς απόψεις κοινωνίας. Συμφωνείτε με αυτές τις δηλώσεις που ανάφερα εδώ περί κοινωνικής οικονομίας. Ε, Κύριε Έτιγκερ, <clears throat> απαντήστε αν θέλετε. Όπως ε, είπατε και εσείς, είναι πολλοί οι τραπεζίτες, κάποιοι τραπεζίτες, οι οποίοι απέτυχαν και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στις υποσχέσεις που είχαν παράσχει σε σχέση με ορισμένα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Ο τραπεζικός τομέας λοιπόν απαιτεί σημαντικές και ε, ριζικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το καθεστώς υποχρεώσεων των ε, τραπεζιτών και των προϊόντων τα οποία παρέχουν. Νομίζω ότι εδώ συμφωνήσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα πρότυπο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των τραπεζικών προϊόντων και την διατήρηση και την δημιουργία δομών για αποζημίωση των καταθετών. Τα πράγματα λοιπόν δεν είναι τα ίδια όπως όταν ήταν πριν από δύο χρόνια. Εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω αυτήν την ε, κρίση και σε άλλες περιπτώσεις. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί οι οποίοι αντίθετα διατηρούν μια κοινωνική αντίληψη του λειτουργήματός τους και δεν θα έπρεπε από ένα κλάδο μονάχα και από ένα τμήμα μονάχα της ευρωπαϊκής οικονομίας να καταλήγουμε σε γενικότερα συμπεράσματα. Αυτό νομίζω θα ήταν λαθασμένο σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα τονίζω και πάλι ότι η κοινωνική οικονομία της αγοράς θα πρέπει να μείνει ο γνώμονας στις δράσεις μας και συγχρόνως να προσθέσουμε και την οικολογική θεώρηση. Κοινωνικά, οικονομικά και οικολογικά θα πρέπει να δούμε τον ενεργειακό τομέα. Σας ευχαριστώ κύριε Έτουγκερ. Απαντήσατε μια πλειάδα ερωτήσεων και όπως προβλέπουν οι κανόνες θα ήθελα να σας δώσω το λόγο εάν το επιθυμείτε να δώσετε τα καταληκτικά σας συμπεράσματα. Έχετε πέντε λεπτά λοιπόν για να το πράξετε αυτό εφόσον επιθυμείτε κύριε Ότιγκερ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για το κλίμα που επικράτησε, το οποίο ήταν, πρέπει να πω, συναρπαστικότερο από ό,τι θα μπορούσα να, να προβλέψω. Ήταν αυστηρή η στάση σας, αλλά δίκαιη και οι ερωτήσεις σας δεν ήταν μόνο, ούτε τις εκλαμβάνω μόνο σε ερωτήσεις, αλλά και ως τοποθετήσεις και τις λαμβάνω υπόψη μου τέτοιες. Έχω την πεποίθηση, έχω την δέσμευση αναλάβει να συνεχίσω τις επαφές μας στη συνεργασία μαζί σας και σε άτυπη μορφή και επισήμως, ε, σε τυπική μορφή στο Στρασβούργο, στις Ολομέλειες και πάντως για λύσεις, για στόχους, για επιφυλάξεις με πάντα διαδεθμένος να συζητώ. Για τον κάθε έναν, για την κάθε μία σας, εδώ είμαι πάντα ανοιχτός και περιμένω να ακούσω τις απόψεις σας. Είστε όλοι εξίσου σημαντικοί για μένα. Οι στόχοι είναι σαφείς, πολλά έχουν ήδη ξεκινήσει και πρέπει να συνεχιστούν, καινούργιοι στόχοι θα προκύψουν και το άρθρο 494 είναι για μένα δέσμευση. Είναι υποχρέωση να εκπληρώσω τα καθήκοντα αυτά που ορίζονται και αυτά θα είναι όσα έχω να κάνω μαζί σας τα επόμενα πέντε χρόνια και μαζί με το Συμβούλιο βεβαίως και κατά την προετοιμασία για την παροχή των υπηρεσιών, όπως οφείλω, και ως εταίρος. Ελπίζω να μου δώσετε να εκδηλώσετε απέναντί μου την εμπιστοσύνη πάνω στην οποία θα μπορούσα να στηριχτώ για να εργαστώ στη δουλειά αυτή και να συνεργαστώ μαζί σας για το μέλλον. Μέσα σε πνεύμα καλό, θετικό, όπως σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ βλέπετε, του κρατηδίου της του Βουστεβέργης, βλέπετε ότι τα χειροκροτήματα δείχνουν, εκδηλώνουν ικανοποίηση για την παρουσία σα εδώ και τι επιδόσει σα. Σταματούμε τη συνεδρία μα εδώ για να συνεχίσουμε το απόγευμα. Έχουμε ακόμη να συζητήσουμε κάποια θέματα των υποψηφίων.